afternoon. Um... yes. Τρεις και τέταρτο αρχίζει ο νομισματικό διάλογος ε, και έχουμε τώρα τη συνήθη να διεκπαιρεώσουμε. Ε, ξέρω ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι είναι λίγο ε, έτσι ακόμα αναστατωμένοι. Καθίστε σας παρακαλώ και κάντε ησυχία. Έγκριση της ημερησίας διάταξης. Μπορούμε να θεωρήσουμε εγκεκριμένη την ημερησία διάταξη. Ωραία έγκριση των πρακτικών της 5ης Σεπτεμβρίου. Να θεωρήσουμε ότι είναι εγκριθέντα και τα πρακτικά. Τα λάβαμε. Ωραία. Μερικές ανακοινώσεις της Προέδρου για να τις διεκπαιρεώσουμε πριν αρχίσει ο νομισματικός διάλογος. Πρώτον, έκθεση ΑΦΚΟ για την πολυεπίπεδη κυβέρνηση πολλαπλών ταχυτήτων. Και θέλω να σας πω για ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και καιρό σχετικά με την έκθεση αυτή επανειλημμένα Έχω εκφράσει τις ανησυχίες της Επιτροπής μας για το πεδίο εφαρμογής αυτής της ε, έκθεσης ε, που αφορά την ε, ΟΝΕ και την Τραπεζική Ένωση που εμείς αυτό το καιρό συζητούμε ή συζητήσαμε στο παρελθόν, είμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων, όπως SSMS, RM, BRD, NTGS και ε, για να σας δώσω μερικά αρχικά. Στις 4 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Κασίνη μου επιβεβαίωσε την ε, προθυμία της Επιτροπής του να εξετάσει ε, τα όσα προτείνει η γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού στο εδάφιο Δέλτα του σχεδίου ψηφίσματος της ΑΦΚΟ. Το εδάφιο Δέλτα καλύπτει ζητήματα αποκλειστικής όμως αρμοδιότητας της Επιτροπής μας και εμείς θα γνωμοδοτήσουμε ε, για να συμπεριληφθεί η γνωμοδότησή μας στην τελική έκθεση της ΑΦΚΟ χωρίς δική τους ψηφοφορία. Εμείς θα ψηφίσουμε, αλλά εκείνοι δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν στη συνταγματική. Επιπλέον, ετελογικές σκέψεις και οι τροπολογίες της ΑΦΚΟ, εκτός του ΔΕΛΤΑ, ε, που μπορεί να μην είναι συμβατές ή συναφείς με τη δική μας γνωμοδότηση που καλύπτει το σημείο Δέλτα και δεν θα πρέπει να τεθούν σε ψηφοφορία. Είχαμε άτυπες συνεννοήσεις, ε, οι συγητές της ΕΚΟΝ και της ΑΦΚΟ. Η ΕΚΟΝ θα ψηφίσει στις 17 Οκτωβρίου τη γνωμοδότηση και είναι μια ημερομηνία που βολεύει και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η έκβαση είναι ικανοποιητική ως προς αυτό. Ε, για τις επόμενες απλουστευμένες διαδικασίες βάσει του άρθρου 46 του κανονισμού οι συντονιστές μας αποφάσισαν στις 10 Σεπτεμβρίου η απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες να ε, εφαρμοστεί στα εξή θέματα. Ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Γαλλίας ε, ως προς τη ε, φορολόγηση των καταθέσεων και διοικητική συνεργασία στο Σαν ε, για θέματα φορολογικής συνεργασίας. Ο κύριος Νίτρας του Έλκη είναι και το δεύτερο είναι μια ε, πρόταση που τροποποιεί τις οδηγίες 2006-112 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2008-118 ε, ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς τις ιδιαίτερα μακρισμένες υπερπόντιες κτίσεις της Γαλλίας, τη Μαγιότ προκειμένου και εισηγητής είναι ο κύριος Κάζα, ενώ η ψηφοφορία θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου. Επίσης θα ψηφίσουμε για μια δεύτερη ε, γρήγορη ε, επίλυση ε, για την οδηγία Omnibus 2 για θέματα φεραγγιότητας 2 το Νοέμβριο θα εγκριθεί στην Ολομέλεια. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα καταθέσει εγκαίρως πράγμα που αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου. Άρθρο 51. Έκον, Λίμπε, το κοινό θέμα αυτό για την οδηγία κατά της νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες και εμβάσματα χρημάτων. Όπως είπαμε, η οδηγία αυτή θα συζητηθεί ε, βάσει του άρθρου 51 συγγνώμη, σε κοινή συνεδρίαση δηλαδή των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕΝ και σε συνεργασία και συνεννόηση με τους τέσσερις συνεισηγητές γιατί είναι δύο να επιτροπή. Ε, ενδεκτικό χρονοδιάγραμμα. Κατάθεση του σχεδίου έκθεσης 6 ε, Νοεμβρίου, τροπολογίες, ε, προθεσμία, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, παρουσίαση των τροπολογιών, υποβολή δηλαδή, 5 Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε Δευτέρα ή Τρίτη 20-21 ε, Ιανουαρίου. Για τους τριμερείς διαλόγους. Ένας τρίτος διάλογος για το μηχανισμό ε, ε, εκαθάριση τραπεζών 18 Σεπτεμβρίου για ένα θεωρημένο κείμενο ε, για τις ειδικέ αρχές και διαχείριση. Έγινε μια πρώτη αλλαγή, ανταλλαγή μάλλον απόψεων σχετικά με τις αρμοδιότητες και αρχές που θα έχει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, EBA. Επόμενος τιμές διάλογος θα γίνει 26 Σεπτεμβρίου και Υπάρχει μια ολόκληρη ανταλλαγή και αλληλογραφία non-paper κατά τα άλλα και ιδεών και κειμένων ε, που κυκλοφορούν δεξιά Λοιπόν, διακοπή ο λίγων λεπτών αφού σας τα είπα όλα αυτά για να αρχίσει ο, τριμερής, ε, ο νομισματικός μάλλον διάλογος. Να ε, πάω να καλωσήσω τον Μάριο και να τον φέρω στην Επιτροπή. Okay, Καλώς λοιπόν θα ξεκινήσουμε αφού βγουν από τη μέση οι φωτογράφοι. Είχα μία μικρή προσωπική ανταλλαγή απόψεων με τον Μάριο και όσοι παρακολουθούν του Twitter θα ακούσετε ότι ζήτησε για ένα για τους Financial Times και όχι μόνο για μια αθλητική εφημερίδα. Δεν ξέρω σε ποια αεροπορική εταιρεία ταξίδευε, αλλά δεν είχανε τους ε, FT, όπως λέει η πρόεδρος, τους Financial Times. Σας καλωσορίζουμε πρόεδρε που θα παρουσιάσετε τις απόψεις της ΕΚΒ για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα και μετά θα περάσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων. Κοιτάξτε, τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ομιλούν για 5 λεπτά. Όσο λιγότερο μιλάτε, τόσο περισσότερες δυνατότητες θα έχετε για να θέσετε και συνοδευτική ερώτηση ή αντερώτηση. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κύριε Ντράγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, είναι χαρά για μένα που σας ξαναγρίσκω. Μετά από τη σημαντική ψηφοφορία της Ολομέλειάς σας για τον κανονισμό SSM του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας, η ψηφοφορία αυτή προ... της ψηφοφορίας αυτής προηγήθηκαν θα έλεγα διαπραγματεύσεις για πάρα πολλά διαθεσμικά θέματα και για τη διαθεσμική συμφωνία, για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σούλτ, την Επιτροπή σας και τη διαπραγματευτική ομάδα μας για την επιτυχή κατάληξη σε σχέση με τον ενιαίο μηχανισμό. Τα δύο θεσμικά μας όργανα μοιράζονται θα έλεγα ένα κοινό συμφέρον για να ολοκληρωθεί δηλαδή το ταχύτερο δυνατόν η ε, Τραπεζική Ένωση. Η συμφωνία αυτή δείχνει και διασφαλίζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας, λογοδοσίας και προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο επικοδομητικό πνεύμα και τους επόμενους μήνες και ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια γρήγορη δημιουργία ε, της ε, Επιτροπής Εποπτείας, του Εποπτικού Συμβουλίου καλύτερα. Θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στον τομέα των οικονομικών και νομισματικό στην περιοχή του ευρώ. Και θα αναφερθώ σε δύο πιο συγκεκριμένα θέματα, τις επιπτώσεις των έκτακτων μέτρων μας και τις νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια της αναθεωρημένης αρχιτεκτονικής της Νομισματικής Ένωσης. Μετά από την συνάντησή μας τον μήνα Ιούλιο πήραμε θετικά στοιχεία για την οικονομία της ζώνης ευρώ. Μετά από έξι τρίμηνα αρνητικής ουσιαστικά ανάπτυξης, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% από τρίμηνο σε τρίμηνο και αναφέρομαι στο δεύτερο του 2013. Τα μέτρα εμπιστοσύνης και κάποια έλεγχη της παραγωγής βοήθησαν, στήριξαν μάλλον αυτούς που πιστεύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα συνεχίσει την αργή της ανάκαμψη και κατά τη διάρκεια του παρόντος τριμήνου παρά τις χαμηλές προβλέψεις στην παραγωγή για τον Ιούλιο. Στο μέλλον η οικονομική δραστηριότητα θα αποφεληθεί. Ε, από μια σταδιακή αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και από την διευκολυντική σε εισαγωγικά πολιτική μας στον τομέα το νομισματικό και από ενισχυμένη ζήτηση για εξαγωγές. Όμως η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή και η ανάκαμψη θα πρέπει να σταθεροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Στον πληθωρισμό ο ετήσιος ρυθμός έπεσε στο 1,3 τον Αύγουστο του 2013, ήταν θυμίζω 1,6 τον μήνα Ιούλιο. Οι υποβόσκουσες πιέσεις στις τιμές θα παραμείνουν ελεγχόμενες και θα αντικατοπτρίζουν την γενικότερη αδυναμία της συνολικής ζήτησης και το αργό βήμα της ανάκαμψης μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για, την, για τον πληθωρισμό συνδέονται με τη σταθερότητα των τιμών. Οι κίνδυνοι θα αντισταθμιστούν τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Η νομισματική δυναμική παραμένει υπό έλεγχο, ο ετήσιος ρυθμός αλλαγής η δανειοδότηση του ιδιωτικού τομέα ε, χαμήλωσε ακόμα περισσότερο, εξασθένησε ακόμα περισσότερο τον Ιούλιο. Αυτό δείχνει το παρόν στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου αλλά και αυξημένους πιστοτικούς κινδύνους στα πλαίσια των ρυθμίσεων ανάμεσα σε αυτούς που δανείζουν και σε αυτούς που δανείζονται. Οι σημαντικές βελτιώσεις στην χρηματοδοτική κατάσταση των τραπεζών από το καλοκαίρι του 2012 δεν έχει τροφοδοτήσει ακόμα περισσότερα δάνεια. Πάνω σε αυτή την εικόνα λοιπόν το Συμβούλιο των Κυβερνητών της Τράπεζας αποφάσισε να συνεχίσει να ασκεί την ίδια πολιτική νομισματική όσο είναι απαραίτητο για να επαναλάβουμε και να επιβεβαιώσουμε αυτήν την υπόσχεσή μας στα πλαίσια μιας σχετικά πτητικής ε, αγοράς νομισματικής. Εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις τον μήνα Ιούλιο ε, λέγοντας ότι τα επιτόκια τα κεντρικά θα πρέπει να παραμείνουν στα παρόντα επίπεδα ή και ακόμα χαμηλότερα για μια ακόμα μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Η προσδοκία αυτή η οποία επιβεβαιώθηκε άλλωστε και τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο βασίζεται σε μια ε, <clears throat> χαμηλή προοπτική για τις πληθωριστικές τάσεις μέσω πρόθεσμα λόγω της ε, γενικότερα ε, ευρείας βάσης αδυναμίας της οικονομίας και των ασθενών γενικά νομισματικών δυναμικών. Θα παραμείνουμε λοιπόν εμείς στα πλαίσια της ε, προσπάθειάς μας για σταθερότητα των τιμών και επίσης για τη σταθεροποίηση της νομισματικής αγοράς. Για να διασφαλίσουμε το σωστό πέρασμα της νομισματικής ε, πολιτικής ε, στις συνθήκες χρηματοδότησης της ευρύτερης οικονομίας, είναι απαραίτητο να πάρουμε μέτρα για να μειώσουμε την πολυδιάσπαση των αγορών των πιστοτικών της ζώνης ευρώ. Η νομισματική πολιτική συνεισφέρει προς την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στις μεταφορές που είπα, εφόσον δεν συνδέονται βέβαια με πιο διαρθρωτικά εμπόδια. Δίδοντας απεριόριστη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από κεντρικής τράπεζες, εφόσον υπάρχει βέβαια κατάλληλες εγγυήσεις, εμείς έχουμε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για να ανακουφίσουμε την πίεση στα πιστοτικά ιδρύματα. Υπήρξε ρύθμιση του πλαισίου ε, των εγγυήσεων έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και τον ισολογισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά να προωθήσουμε επίσης και διαφάνεια ιδιαίτερα ε, στις αγορές των διαθρωμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων οι φερέγγιες τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν με την απαιτούμενη ρευστότητα και θα λειτουργήσουμε ε, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τη μόχλευση που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα κάποια θέματα. Τα OMT, ε, τα οποία ανακοινώσαμε πριν ένα χρόνο, οι οριστικές αυτές νομισματικές συναλλαγές έχουν ε, βοηθήσει έτσι ώστε να αποφευθούν καταστροφικοί κίνδυνοι. Τα OMT ε, είναι πραγματικά ε, μια σημαντική, ένα σημαντικό όπλο στο εσωτερικό της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και προσπαθούν να διατηρήσουν τα κίνητρα για τις κυβερνήσεις έτσι ώστε με τη σειρά τους να διατηρούν δημοσιονομικές πολιτικές φερέγγιες και οι οικονομίες να επανέλθουν σε μια υποστηρίξιμη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών επέστρεψε και η εμπιστοσύνη στη ζώνη ευρώ. Σαν συνέπεια αυτού η διάσπαση των χρηματοδοτικών αγορών στην ζώνη ευρώ έχει μειωθεί κατά πολύ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται όχι μόνο στα έκτακτα μέτρα τα οποία πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και στην προόδο την οποία έκαναν οι κυβερνήσει στα πλαίσια της διακυβέρνησης της περιοχής του ευρώ και μέσω των μεταρρυθμίσεων που ακολουθούν. Οι ροές οι οποίες προβλέπονται, ε, προέρχονται από τις πιεσμένες χώρες έχουν πλέον αντιστραφεί. Έχει διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές των πιστοτικών ιδρυμάτων έχει μειωθεί η εξάρτηση από την χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά αποδεικνύονται και από τις πρόορες επιστροφές ε, δανείων προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είχαν πάρει δάνεια στα πλαίσια των προγραμμάτων αναχρηματοδότησης 2 και 3 ετών. Η αποπληρωμή αυτών των πιστώσεων προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σίγουρα ένα μήνυμα εξομάλυνσης. Αλλά αυτό σημαίνει μείωση και της ρευστότητα που έχουν στη διάθεσή τους τα πιστωτικά αυτά ιδρύματα και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ίδια την αγορά την νομισματική. Θα είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιπτώσεις τις οποίες μπορεί να προκαλέσουν οι εξελίξεις αυτές για το σύνολο της νομισματικής πολιτικής. Τέλος θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια της αναθεωρημένης αρχιτεκτονικής της Νομισματικής Ένωσης. Η αρχιτεκτονική του Μάστριχτ έχει ενισχυθεί ιδιαιτέρως από την αρχή της κρίσης. Η Ευρώπη έχει ενισχύσει την δημοσιονομική και μακροοικονομική της εποπτεία έχει δημιουργήσει μια μόνιμη, ε, ένα μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης των κρίσεων, το ESM, και έχει βελτιώσει επίσης και το θεσμικό της πλαίσιο. Προχωράει γρήγορα προς τον ενιαίο ε, μηχανισμό εποπτείας, το SSM, για τις ε, τράπεζες στη ζώνη ευρώ. Μια βασική προτεραιότητα για το τελευταίο τρίμηνο του 2013 είναι να συμπληρωθεί η προσπάθεια αυτή μέσω του ενιαίου ε, μηχανισμού αξιο, αξιολόγησης ή καλύτερα ανάταξης και εξυγίανσης των τραπεζών. Θέλουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα λοιπόν για τη δημιουργία του μηχανισμού αυτού που θα πρέπει να λειτουργήσει την 1η Ιανουαρίου του 2015, κάτι το οποίο δείχνει ότι το βλέπουμε το θέμα σαν κατεπήγον. Να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις τώρα για τον συγκεκριμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην πορεία προς μια πλήρη νομισματική ένωση. Ήδη από το 2010 και μέσω της αποφασιστικής συνεισφοράς και του δικού σας θεσμικού οργάνου δημιουργήθηκε το ESRB έτσι ώστε να ελέγχονται οι μακροπροληπτικοί κίνδυνοι του πιστοτικού συστήματος στο σύνολό του η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει την γραμματεία του ESRB και στηρίζει συνεπώς ε, τον μηχανισμό αυτό. Ε, φέτος έγινε ένα βήμα επιπλέον μέσω ακριβώς και της δημιουργίας του ε, ενιαίου μηχανισμού εποπτείας του SSM. Το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν θα αναλάβει τις νέες ευθύνες της ανάλογα. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει έτσι ώστε οι νέες αρμοδιότητες να γίνονται με την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και επαγγελματικότητα οι συνέργειες μεταξύ των νέων ε, μηχανισμών εποπτείας και των υπαρχόντων μηχανισμών ε, ε, εποπτείας συνεχίζουν να υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά εμείς θα ξεχωρίσουμε από τη μία την νομισματική πολιτική και από την άλλη τον έλεγχο των πιστοτικών ιδρυμάτων, όπως προβλέπεται στα πλαίσια του κανονισμού SSM. Τόσο ο διαχωρισμός θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να επιδιώκει τη βασική της εντολή που είναι η σταθερότητα των τιμών όπως τον προβλέπει η συνθήκη. Ο πραγματικός διαχωρισμός της νομισματικής πολιτικής και των προβλέψεων για τον έλεγχο των τράπεζων θα εφαρμόζεται και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων αλλά και σε επίπεδο τεχνικού προσωπικού. Θα δημιουργηθεί μια νέα ε, εποπτική επιτροπή η οποία ε, θα συντάξει και θα εφαρμόζει τις αποφάσεις. Ταυτόχρονα οι συζητήσεις του Συμβουλίου των Κυβερνητών θα διαχωριστεί από τις αποφάσεις για τα νομισματικά θέματα. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτές τις δύο αρμόδιότητες θα υπογραμμίζεται άλλωστε και από διαφορετικού τύπου συναντήσεις και συνεδριάσεις. Τέλος, να σας πω κάτι για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα όπως λέμε. Α, ήδη από το 2010 μας ζήτησε το Συμβούλιο να δώσουμε την τεχνική μας εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των ε, προγραμμάτων ε, βοήθειας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΕΛΤΑ Εν τω μεταξύ μας έδωσαν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες και από τη συνθήκη ESM και από την δευτερεύουσα κοινοτική νομοθεσία. Εμείς προσπαθούμε να δράσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσουμε τεχνική βοήθεια επί τη βάση της εμπειρογνωμοσύνης μας, όπως κάναμε και στο παρελθόν Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τις απόψεις μας για την κατάσταση των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξηγούμε ακριβώς τις ε, προτάσεις τις οποίες κάνουμε σαν τμήμα της Τρόικα. Να μην ξεχνάμε όμως ότι το Eurogroup είναι το σώμα το οποίο θα αποφασίσει αν θα δοθεί οικονομική βοήθεια και κάτω από ποιες συνθήκες θα δοθεί η βοήθεια αυτή. Σας ευχαριστώ. Αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και για την προθυμία σας να οδείχνει τόσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε θέματα που αφορούν και την Τρόικα. Είναι θέμα που μας απασχολεί εδώ και μας αφορά στην Επιτροπή μας και δεν μπορούμε βέβαια πάντα δημόσια να το κάνουμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν γίνονται τέτοιε κινήσεις είναι πρόσθεκτες. Πάμε αμέσω στις ερωτήσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Ζαν Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα μπορούσα να σας ε, κάνω ένα, θέσω ένα επίκαιρο ερώτημα, αλλά μάλλον είναι προώρο να σας ρωτάω από τώρα ποιες είναι οι πιθανές ε, επιπτώσεις επανεκλογής της κυρίας Μέρκελ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ε, αλλά ας περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες πρωτού θέσουμε τέτοια ερωτήματα. Ας επανέλθω τώρα στο ρόλο της ΕΚΤ, ε, τον εποπτικό ρόλο της ΕΚΤ. Ε, εκτιμούμε το ότι καταλήξαμε τελικά σε διαθεσμική συμφωνία που κατοχυρώνει μεγαλύτερη διαφάνεια, τηρώντας όμως και τους απαιτούμενους κανόνες περιεχεμήθειας. Ξεκινάει η πιο περίπλοκη περίοδος τώρα, δηλαδή η εφαρμογή όλων αυτών των ε, διατάξεων που έχουν θεσπιστεί. προετοιμάζουμε ένα κοινό εγχειρίδιο, single rule book, ε, για την ενιαία υποπτική αρχή και για την έκτη Μιλήσαμε για το διορισμό του νέου αυτού εποπτικού συμβουλίου. Μας είπατε ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτος ε, διαχωρισμός ανάμεσα στις, στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζα και τον ενδεχόμενο υποπτικό τη ρόλο. Θα ήθελα λοιπόν να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε για την ε, σύνθεση και για το διορισμό των νέων οργάνων, διότι αυτό έχει κέρια σημασία για τη λειτουργία αυτών των νέων θεσμών στη συνέχεια. Σα ευχαριστούμε. Thank you. Um, let me say... Απάντηση Ας θεωρήσω ότι είναι ευρύτερο το ερώτημά σας. Κάντε μία ερώτηση για τα πεπραγμένα, για την προπαρασκευαστική φάση του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού, του SSM. Ε, θα δήλωνα μάλλον σε διότι είναι σταθερή και γοργή η πρόοδος που σημειώνει η ΕΚΤ για να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα βάσει του κανονισμού SSM. Οι εσωτερικές διεργασίες λοιπόν συνεχίζονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέχρι ΔΕ τονώνεται η πρόοδος από τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Έχουμε ειδικέ ε, δομές που μας βοηθούν να προετοιμάσουμε το SSM. Έχουμε ομάδα υψηλού επίπεδου, task force για την εποπτεία ε, Έχουμε ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων επίσης, όπου συμμετέχει φυσικά και η ΕΚΤΕ και όλα αυτά τα όργανα διεξάγουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Για να διευκολύνουμε αυτή τη φάση, 78 ε, άνθρωποι έχουν αποσπαστεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές στην ΕΚΤ αμυστή. Υπάρχουν τέσσερις ε, βασικοί τομείς όπου έχει σημειωθεί πρόοδος. Θα ήθελα να παριθμίσω αρχικά τους τομείς και στη συνέχεια να επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες. Ο πρώτος βασικός τομέας είναι η ανάπτυξη αυτού του Single Rule Book, του κοινού εγχειριδίου. Δεύτερος ε, τομέας είναι η υποβολή αναφορών ε, για τον εποπτικό ρόλο. Τρίτος ε, τομέας είναι ο κανονισμός πλαίσιο για τις εποπτικές λειτουργίες και ο τέταρτος τομέας είναι οι προπαρασκευαστικές εργασίε για τη συνολική αποτίμηση, δηλαδή αξιολόγηση ισολογισμών 130 τραπεζικών ομίλων που αντιστοιχούν στο 85% των στοιχείων ε, τραπεζικού ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στη συνέχεια θα ελέγχονται βάσει του νέου συστήματος. Έχουμε λοιπόν ε, τρεις ε, πυλώνες για την αξιολόγηση των κινδύνων και για τα τεστ κοπόσεως. Θα Ω προ το χρονοδιάγραμμα, θα έλεγα ότι βάσει τη προόδου που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες θα μπορούσαμε ήδη να ε, αποδώσουμε αυτή την πρόοδο στη στενή συνεργασία του ΕΚΤ και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών. Ο μηχανισμός SSM ε, θα αρχίσει να λειτουργεί όπως προβλέπει ο κανονισμός ένα χρόνο μετά την έγκριση του νομοθετήματος. Θα υποβάλουμε αναφορά στο Κοινοβούλιο για την πρόοδο μέσω τριμηνιαίας έκθεσης που θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο Αντόλφο μου λέει ότι μπορεί το Δεκέμβριο να ψηφίσουμε ε, ε, στην Ολομέλεια για το διορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού για να γίνουν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες τώρα η Ελίσσα Φερέιρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω πορτογαλικά, κύριε Ντρέκη. Σάρων, θα μπορούσε να σταματήσει το χρονόμετρο μέχρι να βάλουν όλοι ακουστικά. Σα ευχαριστώ. Ε, Κύριε Ντράγκη, χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλώς ορίζουμε και πάλι. Όπως έλεγαν και οι προλαλήσαντες, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έσωσε το ευρώ με τις ε, απευθείας νομισματικές συναλλαγές. Ταυτόχρονα, όπως είπατε, η έκτη συνδέεται με την ε, Τρόικα. Ε, είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα σε σχέση με την Τρόικα. Στην Πορτογαλία, στη χώρα μου, ε, συμμορφωθήκαμε ως επιτοπλίστων με το μνημόνιο και έχουμε τη διπλάσια σχεδόν ύφεση σε σχέση με τα αρχικώς προβλεφθέντα. Είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η ανεργία ε, και 30% ε, είναι το χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ. Αδυνατούμε να ανοιχτούμε στις αγορές και το δημόσιο χρέος μας υπερβαίνει το 7%. Υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, αλλά αδύναμης και αργής, με την ιδιότητα του μέλους της Τρόικα. Και ε, εφόσον εσείς μεταξύ άλλων δρομολογήσατε τα OMTs, τι θα γίνει, τι έπεται στην Πορτογαλία, τι μπορεί να γίνει. Δεύτερη ερώτηση, σε σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την ιδιότητα του ενιαίου επόπτη. Έχω διάφορες υπερωτήσεις. Πρώτον, ε, για τις νέες λειτουργίες θα ήθελα να σας ρωτήσω θα μπορούσατε να κάνετε την αναθεώρηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών εάν δεν υπάρχει ήδη έτοιμος ο μηχανισμός εξυγίανσης των τραπεζών. Δεύτερη ερώτηση. Εφόσον μιλάμε για το ενίο Ταμείο Εξυγίανσης, γιατί είμαι και συγγήτρια για την έκθεση της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα κοινό δημοσιονομικό απόθεμα, ένα fiscal backstop, ούτως ώστε να έχουμε τουλάχιστον ένα τέτοιο αποθεματικό ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το ε, ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης με το που εγκριθεί, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία του όλου εγχειρήματος. Ε, απάντηση. Ευχαριστώ. Για την ερώτηση που κάνατε για την Πορτογαλία. Όπως είπατε, Βλέπουμε, βλέπουμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Ε, στο δημοσιονομικό μέτωπο είναι σημαντικό και ανέκαθεν το λέγαμε οι χώρες ε, να μην ε, ανερούν όλη την πρόοδο που έχουν σημειώσει για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν νομίζω ότι ήρθε τώρα η στιγμή να μιλήσουμε για διεύρυνση του συστήματος και της χορήγησης πίστης, αλλά ε, εφόσον μιλάμε για δημοσιονομική εξυγένση και το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα πρέπει να τονώνουμε την ανάπτυξη. Δηλαδή ε, πρέπει οι τρέχουσες δαπάνες ε, να μειωθούν και να μειωθεί και η φορολογία. Τρίτον, χρειάζεται πλήρης εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Κάποιες χώρες πρέπει να φέρουν σε πέρας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κυρίως στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών ή άλλες χώρες ως προς τον ανταγωνισμό ή την ανταγωνιστικότητα ή την αγορά εργασίας. Σε πάση περιπτώσει είναι εκ των όνων κάρφ να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Για να διατηρηθεί τώρα η ανάκαμψη στις χώρες. Τι μπορούμε να πούμε. Στην Πορτογαλία υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στον τομέα των ε, αποκρατικοποιήσεων. Αυτό θα πρέπει να το έχετε κατά νου. Όμως, μας δείχνουν οι πρόσφατες εμπειρίες που είχαμε ότι παρότι βλέπουμε ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, ναι, σιγά σιγά μάλλον τα σημάδια μιας οικονομικής ανάκαμψης ε, μπορεί να οδηγήσουν σε βίες αντιδράσεις των αγορών. Είδατε τι έγινε με τα spreads. Ε, με την υποψία ότι μπορεί να γίνει κάτι αρνητικό εκτοξεύονται στα ύψη, βέβαια υποχωρούν στη συνέχεια, αλλά παρόλα αυτά. Η πειθαρχία λοιπόν στην αγορά υπήρχε και θα υπάρχει και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Η δεύτερη ερώτηση ήταν πώς μπορούμε να κάνουμε μία αποτίμηση της ποιότητας ε, των στοιχείων του ενεργετικού εάν δεν λειτουργεί ήδη το ε, SRM, ε, ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι θα έχει δεσπιστεί ο μηχανισμός με το που αναλάβει τα νέα καθήκοντα η ΕΚΤ, οπότε Ε, είναι όντω στενό το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανση, όμως στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό το πρώτο στάδιο θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε κυρίως ή μόνο θα έλεγα εθνικά δημοσιονομικά αποθεματικά για τα στρες τεστ και για τις τριμηνιές αναθεωρήσεις για να παραμείνουμε αξιόπιστοι χρειαζόμαστε εθνικά δημοσιονομικά ε, αποθεματικά θα κάνει η ΕΚΤ την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα τον κάνει και θα καταλήξει συμπεράσματα εάν έχει θεσπιστεί ο μηχανισμός τόσο το καλύτερο, εάν όχι τότε οι εθνικές ε, αρχές ε, θα υπομιστούν την ευθύνη σε ε, μία, όχι το απευκταία μάλλον θα έλεγα κατάσταση, θα υπομιστούν την ευθύνη να αναλάβουν εκείνες αυτό το ρόλο. Τώρα τι γίνεται με τη χρηματοδότηση και τι μπορεί να σταματήσει το SRM η ΕΚΤ θεωρεί ότι αυτή η δεκαετία δεν είναι φιλόδοξη. Ε, το αντίθετο, είναι πάρα πολύ μεγάλη περίοδος και θα συμφωνούσα ότι στο ενδιάμεσο διάστημα θα έπρεπε να υπάρχει μια πιστοτική ε, διευκόλυνση και δεν μιλάμε για μεταφορά πιστώσεων διότι υπάρχει ε, αποκατάσταση, δηλαδή λαμβάνει την πίστη βιομηχανία και την επιστρέφει στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Από τους φιλελευθέρους τώρα η Σιλβί Γκουλά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε και πάλι ενώπιόν μας. Το τελευταίο τμήμα της παρουσίασής σας με προβλημάτισε λίγο. Έχετε την πρόθεση να φύγετε με λαφρά επιδηματάκια από την Τρόικα. Σιγά σιγά. Είπατε τεχνική υποστήριξη, τεχνική συμβουλή, οι συμβουλές που δώσαμε στην Τρόικα και λέτε ότι αποφασίζει το Eurogroup. Και είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα ακριβώς για τους πολίτες. Ποιος αποφασίζει ε, για τα μέτρα της Τρόικας. Εσείς τι είστε ένας απλός σύμβουλος, η Κεντρική Τράπεζα. Η Τρόικα που δεν έχει καμία νομική βάση κατά τα άλλα ως μόρφωμα στις συνθήκες αποφασίζει και αν αποφασίζει το Eurogroup σε ποιο λογοδοτεί παρακαλώ το Eurogroup. Σε ποιο είναι υπόλογο. Απάντηση. Ε, όταν άρχισε η κρίση, όλοι οι παράγοντες, θα έλεγα, ε, πρότειναν να δημιουργηθεί η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, συμμετείχε πλήρως και όσο καλύτερα μπορούσε και έδωσε πραγματογνωμοσύνη και εμπειρογνώμονες και κυβερνήσεις και η δική μας τράπεζα, το Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θεωρήσαμε αυτό μας το ρόλο ότι θα έπρεπε να διαρκέσει όσο διαρκούσε και η κρίση. Μακροπρόθεσμα όμως δεν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να είναι τμήμα της Τρόικα. Να η απάντηση λοιπόν. But in this Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση ποιος αποφασίζει, εγώ τι να πω. Ποιο τι θα πει μακροπρόθεσμα και πότε θα τελειώσει η κρίση και ποιος αποφασίζει, κάποιος άλλος, ε, δεν ε, συμβουλεύεται απρός. Μα κοιτάξτε, δεν αποφασίζει η Τρόικα, το Eurogroup αποφασίζει. Γιατί το Eurogroup αποφασίζει να χρηματοδοτεί τα προγράμματα. Με ε, ε, χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό, από τους φορολογουμένους της κάθε χώρας. Αυτοί καλούνται να πληρώσουν τους φόρους που πηγαίνουν στα προγράμματα. Το Eurogroup είναι ο πολιτικός θεσμός, ας το πούμε, που αποφασίζει για τα προγράμματα. Η Τρόικα έχει μάλλον ρόλο συμβουλευτικό. Και το Eurogroup μπορεί, μπορεί να μην δέχεται συμβουλές, λέει η Πρόεδρος. Προχωρούμε. Θέλετε να επανέλθετε, να ξαναρωτήσετε, Σιλβί, η κυρία Γκουλάρ. Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητώ ε, με τα παιδιά μου, ε, ψάχνω να βρω ποιος στέει για το χάλι του σπιτιού. Ε, και τι λέτε, το Eurogroup, ε, ε, παιδιά τους, αποκαλείται ωραία. Θα τους κολακεύσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Ε, μάλιστα. Ε, σας παραπέμπω και πάλι στο προηγούμενο σχόλιο. Ο Dirk από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην μειώσει ε, τις ποσότητες που ε, διαθέτει στην αγορά περιμένει να ε, δει την πρόοδο για την ποσοτική διευκόλυνση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ε, τριετή δάνεια σε εκατοντάδες ευρωπαϊκές τράπεζες με χαμηλά επιτόκια και χαμηλές εγγυήσεις. Η ε, ομάδα επαφής για τη χρηματαγορά ε, ζήτησε να επανεξεταστεί αυτή η συμφωνία, όπως είπε η Wall Street Journal. Ο κύριος Λίκανεν την περασμένη εβδομάδα σε μια εφημερίδα που γνωρίζετε πολύ καλά, την Κοριέρετε Λασέρα, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, αν χρειαστεί θα δώσει και άλλο μακροπρόθεσμο δάνειο και θα ε, ε, ρίξει χρήματα στην αγορά. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η ομάδα επαφής και τι εννοεί ο κύριος Λίκανεν. Θα προβείτε σε ένα νέο γύρο long term refinancing operation, τέτοιου είδους δάνεια λοιπόν και πότε θα γίνει αυτό για την αναχρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ναι, έχετε δίκιο στην εντύπωσή σας. Να σας πω κάτι όμως για αυτή την αναχρηματοδότηση. Το LTRO στην τριετία από το Σεπτέμβριο του 10 ήταν 331 δισεκατομμύρια επαναπληρωμή που σημαίνει σε 63,5% αντιστοιχεί αυτό ε, ε, της ε, καθαρής εισρωής ρευστών. Ε, στην αγορά από την αρχή λοιπόν της περίοδου. Κοιτάξτε, αυτό που τη μια μπορεί να είναι ένα καλό σημάδι γιατί δείχνει ότι οι τράπεζες εξαρτώνται λιγότερο από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ και μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν είτε μέσω των αγορών, είτε μέσω των καταθέσεων, είτε αλλάζοντας ε, πιστοτικές ε, γραμμές μεταξύ τους. Από την άλλη, οι αγορές παρακολουθούν ε, ε, αυτή τη διαδικασία υπερβολικής ημίρευστότητας και μπορούν να αντιδράσουν βραχυπρόθεσμα ε, αυξάνοντας τα επιτόκια. Εμείς Έχουμε διαφορετικό τρόπο καθοδήγησης και λειτουργίας από ότι το Ηνωμένο Βασιλείο, επωνεί οι Ηνωμένες αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ε, χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και μια περιορισμένη τέτοια αναχρηματοδότηση, LTRO, για να διατηρηθεί βραχυπρόθεσμα η χρηματαγορά ε, στα πλαίσια που εξετάζουμε σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό. Ευχαριστώ. Θέλετε να επανέλθετε με ερώτηση. Όχι. Προχωρούμε. Η πράσινη τώρα. Ο Σφεν Γίγκολτ. Welcome, President. Uh, και εγώ, Πρόεδρε. Λίγες ερωτήσεις για το καθεστώς εφαρμογής του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Καταρχάς ο κανονισμός προβλέπει ένα σαφέστατο διαχωρισμό ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και την εποπτική πολιτική. Εσείς επιβεβαιώσατε με ξεκάθαρο τρόπο τη διάκριση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ με εάν από σήμερα θα υπάρχουν συναντήσεις του μηχανισμού εποπτείας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διαχωρισμός στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Ή θα πρέπει να περιμένετε ε, ώσπου να εγκριθεί ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Δεύτερον, θα υπάρξουν διαφορετικές σταδιοδρομίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έτσι ώστε αυτοί που είναι στην πλευρά της εποπτείας να παίρνουν αποφάσεις τις οποίες δεν θα συμφωνούν, με τις οποίες δεν θα συμφωνούν αυτοί που εργάζονται στο τμήμα της νομισματικής πολιτικής. Τώρα για τα λεγόμενα τεστ των ισολογισμών. Μπορείτε να μας πείτε αν τα κυβερνητικά ομόλογα θα ε, εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας και τέλος θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις των ισολογισμών σε εθνικό επίπεδο δεν θα γίνονται μόνο από εθνικές εποπτικές αρχές αλλά και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα ελέγχουν όχι μόνο θα ελέγχονται όχι μόνο σε ανώτερο επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και το σύνολο των ισολογισμών έτσι ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Να επαναλάβω εδώ ότι η αρχή του διαχωρισμού εφαρμόζεται πλήρως. είναι μια νέα εμπειρία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και τις κεντρικές τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν τις επιμέρους ε, εποπτυχούς ε, ρόλους. Έχουν όμως, ε, έχουμε εμπειρίες ότι οι δύο αυτές αποστολές μπορεί να επιδιωχθούν χωρίς η μία να εισπηδάει στην άλλη θα έλεγα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σας επιβεβαιώσω ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές και από τρίτα μέρη ε, δημοσιονομικούς ελεγκτές. Θα περιμένουμε δηλαδή τη συνεργασία και από ελεγκτικές αρχές άλλων χωρών και επίσης και από ανεξάρτητους συμβούλους του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα για όλες τις χώρες μέλη. Βεβαίως, λέει ο Πρόεδρος. Θα ισχύσει για όλες τις χώρες μέλη. Θα υπάρξει μια σειρά λοιπόν διαγωνισμών καταρχάς, μέσω των οποίων θα επιλογούν οι σύμβουλοι σε εθνικό επίπεδο. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία για επιλογή ενός ε, ιδιωτικού αν θέλετε συμβούλου στο εσωτερικό της τράπεζας. Αυτές οι αξιολογήσεις ε, θα είναι χρήσιμες εφόσον είναι αξιόπιστες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. <coughs> Γιατί αλλιώς θα είναι άχρηστες και αντιπαραγωγικές αυτές οι μορφές ελέγχου. Νομίζω ότι ένα από τα αποτελέσματα που αναμένουμε από τα τεστ αυτά και από την εξέταση των ισολογισμών, την εξέταση των προβλέψεις για κινδύνους κτλ. είναι να διαλύσουμε αν θέλετε αυτή την φαιά εικόνα η οποία επιβαρύνει τον πιστοτικό ευρωπαϊκό τομέα. Ε, η εικόνα αυτή ίσως είναι καρπός και υπερβολικών απόψεων, αλλά το να το λέμε δεν φτάνει. Εμείς απλά θα ρίξουμε φως στον ευρωπαϊκό πιστοτικό τομέα. Έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν. Να πω επίσης ότι το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών είναι εξίσου σημαντικό με την ίδια τη διαδικασία. Γιατί για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη διαδικασία αυτή διαφανή θα πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι ιδιαίτερως διαφανεί. Και όπως είπατε θα πρέπει να αποτραπούν οι συγκρούσεις συμφερόντων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπει την υπόθεση αυτή, όπως επίσης και οι Εθνικές Αρχές Εποπτείας. Αναφέρθηκα πιο πριν στην πολύ καλή σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις εθνικές εποπτικές αρχές. Ε, ρωτήσατε επίσης τι γίνεται και με τα ομόλογα του δημοσίου. Αυτό δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Ε, η ομάδα υψηλού επίπεδου δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα το θέμα. Πάντως ο βασικός μας στόχος να είμαστε απόλυτα αξιόπιστοι. Η ομάδα υψηλού επίπεδου λοιπόν που είναι ε, οι λεγόμενοι εκ των προτέρων επόπτες ε, θα κάνουν μια ανακοίνωση γύρω από αυτό στα μέσα Οκτωβρίου το αργότερο, οπότε όλα αυτά τα θέματα θα διευκρινιστούν. Τώρα για την εποπτική αρχή, το Συμβούλιο Εποπτείας, ε, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αποφασίζει. Το Συμβούλιο αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποφασιστεί ε, από τις αρχές. Δεν έχουν οριστεί ακόμα. Οπότε τι, συνάντηση, τι συνεδρίαση να ζητήσω όταν δεν έχω τα μέλη της ε, αρχής. Μα Εφόσον είναι εκεί τα μέλη και δεν προκυρήσονται, δεν ανακοινώνονται οι συνεδριάσεις, δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, λέει ο κ. Γκίγκολτ. Όχι, κοιτάξτε, η ομάδα υψηλού επίπεδου αποτελείται ίσως από πολλούς από αυτούς που θα είναι τμήμα ε, της ε, Επιτροπής Εποπτείας. Αλλά τα κράτη-μέλη θα το αποφασίσουν και όχι η Κεντρική Τράπεζα. Εδώ επαφιέμεθα στα κράτη-μέλη. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και καλά. Δεν θέλουμε εμείς να παγιδευτούμε από, αυτές, ε, τις, ε, από αυτά τα πολύ σημαντικά θεσμικά ε, βήματα. Πρέπει λοιπόν να, να γίνουν τα βήματα αυτά και όταν γίνουν θα προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, χάσαμε λίγο χρόνο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Θα πρέπει ίσως να καλέσουμε εδώ να έρθει το Eurogroup αν καθυστερεί. Ο κύριος Χουντής. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου έχει σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως μέρος της Τρόικα, θέμα για το οποίο κάνετε και εσείς ορισμένες αναφορές. Πρόσφατα το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της Ελλάδας έφτασε στο επίπεδο του 180% του ΑΕΠ. Αυτό καταρρύπτει αυτή η ανακοίνωση καταρρύπτει τις εκτιμήσεις που έκανε η Τρόικα, της οποίας είσαστε μέλος επαναλαμβάνω, που εκτιμούσε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος ε, θα φτάσει μόλις πρόσφατα στο 175 για να μην θυμίσω παλαιότερες δηλώσεις ότι θα ήταν στο 164. Την ίδια στιγμή το άλλο μέρος της Τρόικα, δηλαδή αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με δημοσιότητα ή με διαρροή εκθέσεων, θέτουν πολλές επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Με βάση αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε και με το γεγονός ότι η Τρόικα, της οποίας μέλος είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επαναλαμβάνω, κάνει τώρα αυτή την περίοδο αξιολογεί την εφαρμογή του προγράμματος και από του ελληνικού προγράμματος και θέλει να αποτιμήσει και το κενό του προγράμματος, σας ερωτώ. Τι λέει λοιπόν η εμπειρογνωμοσύνη του ενός τρίτου της Τρόικα, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Δεύτερη ερώτηση. Συμμερίζεστε την άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι το ελληνικό χρέος πρέπει να πέσει κάτω από το 110% το 2022 για να είναι βιώσιμο. Και το τρίτο, τι συζητάτε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συζητάτε νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Έχετε διαφορετικά σενάρια. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω ότι βασικά αυτό το ερώτημα, αν χρειάζεται και τρίτο πρόγραμμα η Ελλάδα, αυτό είναι, αν χρειάζεται τρίτο πακέτο, αυτό είναι νομίζω πολύ νωρίς να το πούμε, γιατί το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής ε, στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Σκέλος λύγει το τέλος του 2014, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέχρι το 2016 αρχές. Κατά την άποψή μας είναι πολύ νωρίς να συζητήσουμε επιμήκυνση του παρόντος προγράμματος ή παροχή νέου. Και επίσης μια τέτοια απόφαση θα εξαρτηθεί από την πρόσβαση στις αγορές της Ελλάδας στα τέλη του επομένου έτους και είναι πολύ δύσκολο κανείς να το προείπει και να το προβλέψει από τώρα. Ως προς το ρόλο της ΕΚΤ στην Τρόικα, νομίζω το είπα προηγουμένως. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για την νομισματική πολιτική. Και από τη μια σε καιρούς κρίσης είναι καλό που παρέχουμε στην Τρόικα, αλλά δεν δίνουμε ούτε τα προγράμματα, ούτε τη χρηματοδότηση εμείς από την τράπεζα. Ε, δίνουμε ρευστότητα βεβαίως ως υποστήριξη στις τράπεζες και στις ελληνικές αλλά και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, είπαμε ότι ε, θέλουμε εντόνως να είμαστε μέρος της Τρόικας γιατί έτσι βοηθούμε με την εμπειρογνωμοσύνη στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αλλά όπως σας είπα αυτό έχει να κάνει και περιορίζεται στην περίοδο της κρίσης. Δεν έχω να προσθέσω πολλά περισσότερα στα όσα είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Oh, yes, Σύντομα παρακαλώ. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να επανέλθω στο αρχικό μου ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε σε σχέση με ποιε είναι οι σχέσει σα στην Τρόικα με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Επαναλαμβάνω, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο λέει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ότι το ελληνικό χρέο δεν είναι βιώσιμο και προτείνει ορισμένα πράγματα ή ακούγονται ορισμένα πράγματα. Εσεί επ' αυτού θα θέλατε να μου πείτε ποια είναι η δική σα εκτίμηση. Είναι βιώσιμο όταν φτάνει στο 180% το ελληνικό χρέο. Ειλικρινά, η παρούσα ε, ε, θεώρηση είναι ότι είναι βιώσιμο το χρέος και εμείς δεν βλέπουμε κανένα λόγο να το αλλάξουμε αυτό το δεδομένο. Δεν νομίζω να καταφέρετε να σας απαντήσει τίποτα περισσότερο. 100%. 180% από ό,τι φαίνεται είναι βιώσιμο. Ε, δεν ξέρω. Ε, από την EFT, ο Σαν Ποτέρχο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Ντράγκη και να τον καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τη μακροπρόθεσμη πολιτική. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης τα επιτόκια ήταν χαμηλά εδώ και καιρό. Και είπατε ότι θέλετε να συνεχίσετε αυτή την πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ε, όταν αλλάζει τα επιτόκια αντιδρούν οι αγορές. Ε, αν αυξηθεί ας πούμε το κατευθυντήριο επιτόκιο έστω και ελάχιστα ε, αναστατώνονται οι αγορές και θέλω να σας ρωτήσω αυτή η κατάσταση που επικρατεί αυτό τον καιρό θεωρείται φυσιολογική την αντιλαμβάνονται έτσι οι αγορές και πότε ε, υπολογίζεται να μπορούν να αυξηθούν τα επιτόκια και μακροπρόθεσμα, γιατί ανησυχούμε πολύ εμείς, διότι ε, όταν είναι χαμηλά τα επιτόκια ευνοείται ε, ο δανεισμός, ενώ οι χώρες δεν θέλουν να προωθούν το δανεισμό, οι χώρες μας τουλάχιστον. Ευχαριστώ οι επίσημες κατευθυντήριες γραμμές λένε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τωρινό ή χαμηλότερο επίπεδο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Αυτή η βασική και επίσημη κατευθυντήρια γραμμή εδράζεται επί της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του πληθωρισμού. Σας είπα τον Αύγουστο για την περιζώνη ευρώ από 1,6 τον Ιούλιο έπεσε στο 1,3 ε, και προσδοκάται πως θα παραμείνει κάτω του 2% πιο κοντά στο 1% παρά στο 2% για παρατεταμένη χρονική περίοδο, όπως σας είπα. Και δεδομένης της αδυναμίας ε, της οικονομίας ε, και της υψηλής ε, ανεργίας. Αυτή είναι η μεσοπρόθεσμη αποτίμηση και ως εκ τούτου η νομισματική μας πολιτική που εντολή έχει να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών προς τις δύο κατευθύνσεις, προς τα κάτω και προς τα πάνω έχει εκδώσει αυτή την επίσημη κατευθυντήρια γραμμή. Οπότε Ξαναλέω, αναμένεται τα επιτόκια να παραμείνουν στα τωρινά και χαμηλότερα επίπεδα για μεγάλη χρονική περίοδο. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες περιπληθωρισμού ε, εξακολουθούν να ε, βασίζονται στα οικονομικά στοιχεία που έχουμε και άρα θα πρέπει να έρθουμε ε, να έρθουμε αντιμέτωποι με νέα ενδεχομένω οικονομικά σενάρια. Αλλιώ θα παραμείνει η κατάσταση ω έχει για μεγάλη χρονική περίοδο όπω σα είπα. Ε, και αυτό που κρύβεται κατά πάσα πιθανότητα πίσω από το ερώτημά σα, είναι το εξή ότι αληθεύει ότι τα επιτόκια, ε, αν παραμείνουν χαμηλά για μεγάλη ε, χρονική περίοδο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερου κινδύνου και το έχουμε βιώσει αυτό στο παρελθόν. Όμω, Πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι πλήρως για τους κινδύνους για την νομισματική σταθερότητα που μπορεί να προκύψουν από τα χαμηλά επιτόκια και θα χρησιμοποιήσουμε τη αυτή περίπτωση, μακροπροληπτικά εργαλεία. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Προς το παρόν είναι ισχνές οι ενδείξεις που έχουμε ότι κάτι τέτοιο σημαίνει. Ευχαριστώ. Uh, Χαίρομαι που αναφέρθηκατε στη μακροπολιτική εποπτεία, θα επανέλθουμε σε αυτό. Δεν ξέρω, θέλετε συμπροματική ερώτηση ή όχι. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Βέρνε Λάγκερ, ο οποίος λάμπει. Äh, ναι, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τώρα υποστήριζα μαζικά τα μέτρα της ΕΚΤ και υπό την έννοια ότι είστε το μόνο θεσμικό όργανο στην κρίση που είχατε τη δυνατότητα να δράσετε. Γι' αυτό θα ήθελα να διαφωνήσω με τους συναδέλφους που θέτουν και πάλι πρόβλημα τρόικα εδώ για δέκατη ή δωδέκατη φορά. Εγώ το θεωρώ πολύ απαραίτητο να συμμετέχετε εκεί. Αλλά δεν συμφωνώ με όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό θα ήθελα και σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Γκίγκολτ να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις ε, για το διαχωρισμό της νομισματικής πολιτικής με την εποπτεία. Αυτό είναι σημαντικό. Είπατε και δηλώσατε βέβαια ότι θα υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός στην νομισματική πολιτική, είστε ανεξάρτητοι μεν, στην εποπτεία χρειάζεστε και εσείς έλεγχο. Θέλετε και εσείς τον έλεγχό σας, είτε από κυβερνήσεις είτε από κοινοβούλια. Όλες οι εποπτικές αρχές πρέπει να ελέγχονται με τη σειρά τους. Ποιος θα είναι ο ελεγκτής, γιατί υπάρχουν και προβλήματα ε, και μάλιστα στο στήσιμο του μηχανισμού η συνάδελφος πρόεδρος είπε το Δεκέμβριο θα αποφασίσουμε διορισμό πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Αλλά πρέπει να αρχίσετε από τώρα να στείνετε αυτό το όργανο. Οι εθνικές ελεγκτικές αρχές πώς θα συμμετέχουν σε αυτή τη φάση την αρχική της εποπτείας. Έχω και άλλη ερώτηση. Τι γίνεται με το Ταμείο Εξυγίανσης που σωστά ζητάτε από την 1η του 2015 να λειτουργεί. Τι απαντάτε στον κύριο Άσμουσεν να χρησιμοποιείται μέχρι τότε ο μηχανισμός σταθερότητας ESM και ε, ακόμα και το ταμείο αυτό να εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με αυτό δεν το θεωρείτε επικίνδυνη συγκέντρωση εξουσίας και τα νομισματικά και τα εποπτικά και μήπως χαθεί έτσι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ε, για την νομισματική πολιτική μια άλλη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ιαπωνική τυπώνουν μαζικά χρήμα και, πέφτει και το, πέφτουν και τα επιτόκια στο Το είπατε κι εσείς ότι είναι επικίνδυνο αυτό για τα συνταξιωτικά συστήματα, για ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και τη χαρακτηρίζουν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απλώς αυτό θα το σημειώσει και θα λάβει γνώση ή θα προσπαθήσετε διεθνώς να πιέσετε για μια μετριοπαθή ε, πολιτική στραμμένη προς τα επιτόκια. Thank you. Um, Ναι. Καλό θα ήταν να έχουμε έτοιμο το Ταμείο Εξυγίανσης που θεσπίσαμε, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί να μην χρειαστούμε 10 χρόνια, αλλά να είναι συντομότερος ο χρονικός ορίζοντας. Εντάξει. Και σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σας πως ε, η ΕΚΤΕ καμία δουλειά δεν θα έπρεπε να έχει με αυτό το Ταμείο. Δεν ξέρω αν πέρασε από το μυαλό κανενός εδώ μέσα ότι η ΕΚΤ θα έχει κάποια σχέση με το Ταμείο. Δεν θα έπρεπε και δεν θα έχει καμία σχέση. Αληθεύει επίσης ότι όσο υποχρηματοδοτείται το Ταμείο θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού για το Ταμείο από κάποια άλλη πηγή. Και εδώ ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα ε, εναλλακτικών λύσεων και ούτω ή άλλω είμαστε πρόωρο στάδιο προβληματισμού. Κάποιοι είπαν ότι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα θα μπορούσε να δώσει αυτό το Ταμείο Εξυγίανση σε μία πιστοτική γραμμή. Δεν είμαι σίγουρο ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο δυνάμει τη ισχύουσα συνθήκη, αλλά ε, σίγουρα είναι υπαρκτό το πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί τρόπον κοινά. Για το δεύτερο ε, ε, ζήτημα. Με ρωτήσατε για το Εποπτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δουλειά της ΕΚΤ να διορίζει οποιονδήποτε. Τα κράτη-μέλη έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Όταν γίνει ο διορισμός του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών, συγγνώμη, του Εποπτικού Συμβουλίου, τότε ε, θα μπορέσουν να διεξαχθούν και οι συνεδριάσεις αυτού του Συμβουλίου. Για τα χαμηλά επιτόκια που μου είπατε, κατανοώ τις ανησυχίες που εκφράζεται για τους κινδύνους που δημιουργούν τα χαμηλά επιτόκια, όχι μόνο για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως σας έλεγα προηγουμένως, αλλά για τις ε, ασφάλειες, ασφάλειες ζωής, ε, συντάξεις, ε, αλλά και γενικότερα για τους καταθέτες, για όσους έχουν αποταμιεύσει και βλέπουν να τιμωρούνται λόγω μιας παρατεταμένης χρονικής περίοδου χαμηλών επιτοκίων. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια νομισματική πολιτική για το σύνολο της Ευρωζώνης. Αυτή είναι μια απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Δεύτερον, δείτε τη συμπεριφορά των επιτοκιών κυρίως στη Γερμανία το τελευταίο τρίμηνο ή τετράμινο. Αυξήθηκαν παρότι τα δικά μας τα επιτόκια έχουν παραμείνει ίδια. Ο λόγος ποιος είναι για τα ε, κυβερνητικά, τα δημόσια ομόλογα ήταν τεχνητά χαμηλά τα επιτόκια, διότι ήταν ένας ε, παράδεισος κεφαλαιακών ροών η Γερμανία από την υπόλοιπη ε, Ευρωζώνη. Τώρα όμως που ανακτά την εμπιστοσύνη, αυτές οι ροές δεν είναι τόσο ισχυρές όσο στο παρελθόν και βλέπετε ότι και άλλες διεθνές ροές μπορούν να έχουν το ευκταίο αποτέλεσμα, αύξηση δηλαδή των κεφαλαιακών ροών για τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας. Τώρα, περί, ε, από καιρού εις καιρών συζητούμε ε, με τους συναδέλφους ανά τον κόσμο όμως δεν φτάνουμε στο επίπεδο του συντονισμού. Υπάρχει μια ανταλλαγή πληροφοριών σε αυτές τις συζητήσεις, γίνονται συζητήσεις και για ζητήματα που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική σταθερότητα σίγουρα γίνονται τέτοια συζητήσεις, αλλά δεν φτάνουν τον συντονισμό. Σας ευχαριστούμε, Παύο Ζέλμπα, ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε αγαπητέ Πρόεδρε Τράγκη. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι θετικά τα μηνύματα και τα σημάδια ανάκαμψης Ακόμη και η κυρία Φερέιδρα το αναγνώρισε για την Πορτογαλία. Συμφωνώ επίσης με αυτό που είπατε την περασμένη εβδομάδα, ότι η Τραπεζική Ένωση θα βοηθήσει και θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει όμως να έχουμε επίγνωση το γεγονότος ότι αυτά τα θέματα είναι μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βράχει πρόθεσμα, όπως πολύ καλά είπατε, οι πιστώσεις και ε, κυρίως οι ε, χορηγήσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν προβληματικές. Και μένα με ανησυχούν τα χαμηλά επιτόκια, όπως είπε ο κύριος Λάγκεν, αλλά για άλλους λόγους, γιατί δεν έχει αυτό επίπτωση στις χώρες μας. Ε, στη χώρα μου έχουν πρόβλημα χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 25% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το πρώτο πρόβλημα και για τις υπόλοιπες είναι. Και αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν πληρώνουν πενταπλάσια επιτόκια από τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες εταιρείε στην Ευρώπη. Ο κύριος Έππινγκ αναφέρθηκε στα όσα δήλωσε ο κύριος Λίκανεν ότι είστε έτοιμοι να διοχετεύσετε ρευστότητα στην αγορά. Αν γίνει αυτό, αν γίνουν αυτές οι νέες ενέσεις ρευστού, εσείς πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι η ρευστότητα αυτή θα φτάσει στην πραγματική οικονομία στις χώρες μας και δεν θα αναλωθεί σε μέγα τμήμα να χρηματοδοτήσει την αγορά δημοσίου χρέους. Επαναλαμβάνω και επιμένω πώς θα εξασφαλίσει τη ρευστότητα αυτή να φτάσει στην πραγματική οικονομία. Αν ρίξετε λοιπόν φρέσκο χρήμα στην αγορά σε θα φτάσει στις επιχειρήσεις αυτό ή θα αναλωθεί στο δημόσιο χρέος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Let me first agree with you that... Uh, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω μαζί σας ότι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως στις χώρες που επλήγησαν βαθύτατα από την κρίση. Θα συμφωνήσω επίσης μαζί σας όταν λέτε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης αυξήθηκαν τα προσκόμματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Εν μέρη αυτά τα προσκόμματα προκύπτουν από την επιδείνωση της δικής τους οικονομικής κατάστασης. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πολύ υψηλή μόχλευση σε κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή το εφιστάμενο χρέος είναι ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ε, φυσικά ε, ε, επισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Ο ένας είναι η αποτροπή, η αποφυγή μάλλον του κινδύνου, risk aversion από τις τράπεζες. Δηλαδή ακολουθούν πολιτική δανεισμού στου στους κινδύνους σε πολλές χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση. Όμως το επίπεδο δεν είναι αρκετά υψηλό για τις τράπεζες για να συνεχίσουν να δανείζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όπως σας είπατε, όπως είπατε και εσείς, αντί να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, οικονομία επαναγοράζουν κρατικό χρέος. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά και θεωρούμε ότι περισχύει αυτή η τάση. Δηλαδή όντως οι ισολογισμοί των ΜΜΕ είναι σε αδύναμη κατάσταση. Αποφεύγουν τους κινδύνους οι τράπεζες αλλά ένας άλλος λόγος είναι η έλλειψη ζήτηση. Και έγινε μία έρευνα στις επιστοτικές δροές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δύο κάνουμε έρευνες βασικά. Τη μία με τις τράπεζες και ρωτάμε τις τράπεζες γιατί δεν δανείζετε τις μικρομεσαίες. Ε, και μία άλλη που δεν γίνεται τόσο συχνά είναι μία έρευνα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ρωτάμε τις μικρομεσαίες γιατί δεν δανείζεστε εσείς. Ο πρώτος ε, λόγος ε, μη που αναφέρουν είναι η έλλειψη πελατών. Και ο δεύτερος, έλλειψη ε, πιστοτικού αποθέματος. Οι κεφαλαιοκές ροές λοιπόν παραμένουν σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω της έλλειψης πελατών, έλλειψης ζήτησης. Εάν συχνά ε, κάποιοι κάνουν ένα παραλληλισμό με το Funding for Lending, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε ένα ευρύ φάσμα αντισυμβαλωμένων με μια μεγαλύτερη ποικιλία εγγυήσεων και μακρά ορίμανση. Αυτές είναι οι τρεις συνιστώσεις αυτού του Βρετανικού προγράμματος και το ίδιο ισχύει και για τις δικές μας τις ε, επιχειρήσεις αναχρηματοδότησης, μακροπρόθεσμη επιχειρήσεις αναχρηματοδότησης LTROs και αυτό ισχύει μέχρι τέλος του 2011. Έχουμε αναλάβει πολλαπλά μέτρα και πιο πρόσφατα αποφασίσαμε ότι θα μειώσουμε τις απαιτήσει ε, για, ε, για κάποια ε, είδη ενεργητικού, κυρίως αυτά που χρησιμοποιούνται για το δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, μειώσαμε τις αξιώσεις, δηλαδή μπορού, μπορεί η αξίωση να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση όταν η ίδια η τράπεζα θα πάει να δανειστεί από την έκτη για να δανείσει στη συνέχεια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, όταν ε, συζητήσαμε, σε μία από αυτές τις περιοδικές συζητήσεις ε, που κάνουμε για αυτό το ζήτημα, μιλήσαμε και για το ε, πάγιο σύστημα εγγύσεων και εκεί συζητήθηκε το ζήτημα των εγγύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και μιλήσαμε για αυτό το θέμα των αξιώσεων που θα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέρα από την πιστοληπτική ικανότητα που απαιτεί η έκτη για το δανεισμό. Τώρα, κατά την ανοικοδόμηση του συστήματος ε, κύριο μέλημά μας είναι υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς το παρόν σε σχέση με τις μικρομεσαίες είναι αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό ο ρόλος μας προς το παρόν. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος ότι παρά είναι ε, μεγάλες ερωτήσεις. Αν υποδηματά τώρα. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θα μείνω σε αυτό το θέμα με τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Έχω και εγώ διαφορετικές ανησυχίες από αυτές του συναδέλφου Λάγκελ. Ο συνάδελφος Ζάλμπα μίλησε για την κατάσταση στην ε, Ισπανία. Εγώ θέλω να σας πω ότι σε αντίθεση με, τους, με τις ανησυχίες του συναδέλφου Λάγκελ, σε πολλές χώρες υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας και υπάρχουν τεράστιες αποκλήσει στα επιτόκια δανεισμού μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Στη Γερμανία οι επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν με ένα επιτόκιο γύρω στο 1%. Στη χώρα μου και σε άλλες χώρες οι επιχειρήσεις δανείζονται όταν βρουν χρηματοδότηση με επιτόκια κοντά στο 7% και το 8%. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση, συνάδελφε. Ε, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι τον τελευταίο χρόνο τρεις από τις μεγαλύτερες, γιατί μιλήσαμε πριν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τρεις από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό για να βρουν χρηματοδότηση και τελευταίο παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, η Βιοχάλκο, ο μεγαλύτερος μεταλλουργικός όμιλος, μετέφερε την έδρα του στο Βέλγιο για να μπορέσει να δανειστεί. Επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνδέεται ευθέως με αυτό που είπατε, την ομαλή μεταφορά της νομισματικής πολιτικής. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, ούτε ισπανικό, ούτε πορτογαλικό. Θέλω να σας ρωτήσω τι μέτρα ε, ε, μπορείτε και αν σκοπεύετε να πάρετε για να μην φτάσουμε να θεσμοθετήσουμε δύο ταχύτητες στην Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, λοιπόν, ας προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα για το πώς είναι σήμερα αυτός ο κατακαιρματισμός. Στην αρχή της κρίσης υπήρχαμε κατέρωθεν κατακαιρματισμό και στην χρηματοδότηση και στη δανειοδότηση ε, και στην λήψη δανείων. Δηλαδή, είχαμε τις χώρες που είχαν ε, κόστος χρηματοδότησης πολύ περισσότερο χώρες περιφέρειες σε σχέση με τις χώρες του κέντρου και η ρευστότητα ήταν πολύ χαμηλότερη σε χώρες υποποίηση σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ξεπεραστεί. Αυτό που είδαμε τους τελευταίους έξι μήνες θα έλεγα είναι το εξής οι καταθέσεις, με την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης, οι εσωτερικές καταθέσεις επέστρεψαν στις εγχώριες τράπεζες. Και εκεί τι κάνουμε, κοιτούμε την μεταβολή, την αύξηση των καταθέσεων σε κάθε χώρα. Ε, έχουμε ένα συντελεστή διασποράς ε, κατακαιρματισμού μεταξύ ε, των διαφόρων συντελεστών των καταθέσεων τώρα είναι στο ίδιο επίπεδο ε, με το 2007 οι δείκτες αυτοί. Λοιπόν, συμπέρασμα. Η χρηματοδότηση μέσω του κερματισμού των καταθέσεων σε μεγάλο βαθμό έχει εξαφανιστεί. Τώρα, οι αγορές όταν πρέπει να προσφεύγουν στις ε, αγορές και να ε, εκδίδουν ε, ομόλογα και χρέος. Πραγματικά εκεί υπάρχει μια διαφορά και σε σχέση με τα spread. Τώρα, στην δανειοδότηση ε, των επιχειρήσεων μπορεί να υπάρχει διαφορά σε διάφορα σημεία της Ευρωζώνης. Είναι ακόμα διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούν και υπάρχουν και αποχρόντες λόγοι γι' αυτό. Αν κοιτάξτε ε, το... τα ασφάλιστα κινδύνου μιας ε, χώρας υποπίεση και μιας χώρας που δεν είναι υποπίεση υπάρχει φυσικά μια μεγάλη διαφορά. Ε, τα κρατικά ομόλογα επίσης έχουν διαφορετικά επιτόκια. Ε, και κάποιος προλαλής σας αναφέρθηκε σε αυτό. Πολύ συχνά οι τράπεζες αντί να δανείζουν την πραγματική οικονομία αγοράζουν κρατικά ομόλογα που έχουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο και μια απόδοση που τους ικανοποιεί για την καρδοφορία τους. Ε, υπάρχουν τέτοια ζητήματα αλλά και πάλι ο βασικός λόγος είναι η ζήτηση βλέπουμε ότι σταδιακά ε, η νομισματική μας πολιτική μεταφέρεται στην οικονομία και σιγά σιγά ανακάμπτει το σύστημα. Όσο συνεχίζεται αυτή η ανακάμψη μπορεί να δούμε κατακαιρματισμό και να μειώνεται μάλλον αυτός ο κατακαιρματισμός και στο δανεισμό των τραπεζών και θα είναι λιγότερο επισφαλές να δανείζει κανείς επιχειρήσεις. Ναι, αν ήταν μηδενικό ο κίνδυνο των κρατικών ομολόγων, ε, ε θα πηγαίνανε να δανείσουν τι επιχειρήσει αντί να αγοράζουν κρατικά ομόλογα οι τράπεζε. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Λούλινγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφός σας και συμπατριώτης μου, ο κύριος Μέρσος από το Διευθυντήριο της Κεντρικής Τράπεζας, που με την εμπειρία του βοηθά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από τα προβλήματα που είχε έτσι ώστε να μπει στο Διευθυντήριο, έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις στον τύπο. σχετικά με τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, το SSM, που αφορά καταρχάς 130 τράπεζες. Το πρώτο στάδιο θα τεθεί σε λειτουργία σε μια κοντινή χρονικά φάση. Παραμένει όμως το θέμα του backstop, λέει η κυρία Λούλινγκ. Δηλαδή, πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κατανομή των ανακεφαλαιοποιήσεων που θα κριθούν ότι είναι απαραίτητες ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες εφόσον υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στον προϋπολογισμό ενός πιστοτικού ιδρύματος. Θα ήθελα με κάποιο τρόπο να μας εξηγήσετε εδώ ακριβώς τι παίζεται. σχετικά με το Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο είναι υποσυζήτηση, ή Ταμείο Ανάταξης. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Θα ήθελα να προσπαθήσετε να μου δώσετε εξηγήσει για τη διάρθρωση ανάμεσα στην λογική του backstop από τη μία και στο Ταμείο Εξυγίανσης το SRM από την άλλη. Υπάρχει μια συμπληρωματικότητα, πρόκειται για το ίδιο πράγμα ή πρόκειται για δύο πράγματα εντελώς αντιθετικά μεταξύ τους. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε, ο οικονομικός δημοσιογράφος Longley εξηγεί ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αρχίσει και υποχωρεί πλέον και παρουσιάζει σαν απόδειξη το ότι οι ροές διεθνών κεφαλαίων ε, μειώνονται με πολύ σημαντικό τρόπο, ιδιαίτερα στη ζώνη ευρώ από το 2008 και μετά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν και εφόσον αυτό το ε, φαινόμενο επιβεβαιούται, η μείωση των κεφαλουχικών διεθνών ροών, ιδιαίτερα στη ζώνη ευρώ, είναι πρόβλημα αυτού ιδιαίτερα για τη διαχείριση του ενιαίου μας νομίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτησή σας. Εμείς δεν βλέπουμε να αμείωται η παγκοσμιοποίηση. Αν δείτε το τι συμβαίνει με τις ροές των κεφαλαίων από την αρχή του χρόνου και μετά και επίτα θα δείτε ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι ροές των κεφαλαίων συνεχίζουν περαδόθε, ταξιδεύουν τα κεφάλαια ελεύθερα δημιουργούν διαφορετικές νομισματικές συνθήκες, αλλάζουν πολλές φορές τα επιτόκια και σε σχέση επίσης με την αλλαγή ε, από το ένα νόμισμα στο άλλο. Εν πάση περιπτώσει Before you massive flows υπάρχουν δυνατότητες σε ορισμένες περιπτώσεις παρέμβασης, σε άλλες όχι. Υπάρχουν ροές, συνεχίζουν οι ροές και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν υπάρχουν δυνατότητες υπάρχουν έξοδοι κεφαλαίων από παρθένες αγορές που δεν έχουν επηρεάσει αρνητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ροές των κεφαλαίων παραμένουν, είναι κινητικές και η παγκοσμιοποίηση παραμένει όπως την γνωρίζαμε. Τώρα για το SRM, τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, στα πλαίσια της διαβούλευσης εξεφράστης στις αρχές του μήνα. Η επίσημη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα, ε, θα δημοσιευθεί τάχιστα. Το SRM, ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας για την εποπτεία και την εξυγίανση, όπως λέει η απόφαση του Συμβουλίου για να λειτουργήσει σωστά η χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν περιμένουμε τις αποφάσεις του SRM που έχει ένα ενιαίο μηχανισμό, μια ενιαία αρχή και ένα ενιαίο ταμείο. Υποστηρίζουμε λοιπόν και την προβλεπόμενη, ε, τις προβλεπόμενες χρονικές προθεσμίες για τη λειτουργία του SRM από το 2015 και μετά. Σχετικά τώρα με τους δύο τρόπους αξιολόγησης της βιωσιμότητας μιας τράπεζας και ένα πράγμα που θα κρίνει δηλαδή το τι θα κάνει η τράπεζα και από την άλλη το ποιος θα αναλάβει το τι θα γίνει. Το ένα θα το κάνει φυσικά ο μηχανισμός εποπτείας, το άλλο μάλλον θα το κάνει ο SRM. Λοιπόν, γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι η παρουσία της θα πρέπει να είναι παρουσία παρατηρητή. Σε επίπεδο νομικής βάσης τώρα, από ό,τι μας πληροφόρησαν οι νομικές μας υπηρεσίες, το 141 της συνθήκης είναι η κατάλληλη πιθανή νομική βάση για τον κανονισμό λειτουργίας του SRM, του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Η άποψη αυτή ισχύει και για τις νομικές υπηρεσίες και των ε, ευρωπαϊκών οργάνων, θεσμικών οργάνων γενικότερα. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου μας είπε ότι το 114 μάλλον λέει ο Πρόεδρος είναι επαρκές. Τώρα για το λεγόμενο backstop. Χρησιμοποιείται ο όρος αυτός για πολλούς <clears throat> λόγους. Αυτό που λέμε εμείς backstop στο πλαίσιο του SRM είναι το ότι το ταμείο που θα δημιουργηθεί, το ενιαίο ταμείο που θα ελέγχεται από το SRM, χρειάζεται 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί, για να συμπληρωθεί. Οπότε τι θα γίνει αν πριν το τέλος της δεκαετίας υπάρξει πραγματική ανάγκη για τη χρήση του συγκεκριμένου ταμείου. Η δυνατότητα για το ταμείο αυτό να δανειστεί χρήματα, όχι δωρεάν, να δανειστεί από άλλους χρήματα είναι μια δυνατότητα η οποία συζητιέται και η οποία ονομάζεται backstop. Η δυνατότητα δηλαδή να έχει το SRM μια γραμμή πίστοσης από την οποία να μπορεί να παίρνει χρήμα εφόσον δεν έχει αρκετά χρήματα στο εσωτερικό του ταμείου. Ευχαριστώ. Η Έμιλη από Σοσιαλιστές και Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με αυτά που είπατε για τις σχέσεις σας με άλλες κεντρικές τράπεζες. Πολύ ενδιαφέρον. Είπατε ότι κάνετε συζητήσεις αλλά τίποτα επίσημο, καμία δομή λήψης αποφάσεων. Ε, αυτό είναι ε, μεγάλο ελάττωμα του συγγυρίσματος που κάνουμε μετά την κρίση. Δηλαδή, ε, δεν, ποια είναι η θέση μας στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική. Αυτό είναι ένα μόνο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Ε, ας περάσω σε ερωτήσεις. Μιλήσαμε για τον εποπτικό ρόλο της ΕΚΤ και... Οι συνάδελφοι έκαναν την ίδια ερώτηση αλλά δεν πήραν ικανοποιητική απάντηση για την ε, το review, την έκθεση. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο κύριος Δέσσεμπλουμ είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται με ποιοτικό τρόπο η αποτίμηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και εσείς μιλήσατε για αξιοπιστία. Πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως, δεν είχε συγκεκριμένε προτάσει σε σχέση με το πώ θα το κατοχυρώσουμε αυτό. Όχι μόνο την ποιότητα τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, αλλά και πώ θα κατοχυρωθεί η ε, ανεξαρτησία, μεροληψία των εμπειρογνωμόνων. Υπό το φως των επικρίσεων μετά το τελευταίο τεστ κοπόσεως που έγινε και τις επικρίσεις που ακούσαμε για τις μεθόδους, τι έχετε να προσθέσετε και όταν μιλάμε για τους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα, πώς ορίζετε εσείς τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Ε, μιλήσατε για τα backstops, τα ε, δημοσιονομικά αποθεματικά και είπατε ότι πρέπει σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν, ρωτώ εγώ, είναι ρεαλιστικό να ζητάμε κάτι τέτοιο για την Ισπανία, για την Ελλάδα ή ακόμη και για τη Γαλλία. Θα ήθελα να πω ότι η πλήρης αξιολόγηση θα βασίζεται σε μία πολύ σχολαστική και πλήρη μεθοδολογία που τώρα προετοιμάζουμε στα πλαίσια των γενικότερων προεργασιών για τη ε, θέση σε λειτουργία του SSM. Σας είπα ότι θα βασιστούμε στην εμπειρία πεπειραμένων εξωτερικών συνεργατών και έχει κάνει πρόταση υποβολής προσφορών η ΕΚΤ και έχει ήδη προσλάβει εξωτερικό σύμβουλο. Δεύτερον, ε, για, ε, θα έχουμε μία μονάδα που ε, θα τη διαχειριζόμαστε κέντρικα για τα projects με στόχο να εφαρμόζεται αυτή η μεθοδολογία με ανεξαρτησία και ισοτιμία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα υπάρχει συνοχή ε, και αμεροληψία στην εφαρμογή της ε, μεθοδολογίας ε, και θα, δίν, θα ελέγχεται κεντρικά. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε φάμιλα αποτελέσματα της αποτίμησης και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε εξωτερικούς συνεργάτες για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα. Θα συνδέσουμε τις προσπέθειες μας με την κατοχήρωση της ποιότητας της μεθοδολογίας. Μόνο έτσι θα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Για τα αποθεματικά... Λάβαμε υπόψη ότι έχουν πολύ, μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερα αποθεματικά ούτως ή άλλως οι τράπεζες μετά την κρίση και άρα είναι ρεαλιστικό να έχουμε τέτοια εθνικά αποθεματικά ακόμη και για τις χώρες ε, τις οποίες αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Έμιλι, ο Υπουργός Ντάισελμπλουμ ήταν ε, απόλυτος ε, και για την ιεραρχία και για τη χρήση εμπειρογνωμόνων και παροχή συμβουλών. Ε, νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφή στις δηλώσεις του. Λοιπόν, τώρα που πάω στο Έλκα και τη Μαριάν Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πω Ολλανδικά. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την παρουσία του εδώ ενώπιόν μας. Έχω τις εξής επιφυλάξεις αλλά και το εξής ερώτημα κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καλύψει όλα τα θεσμικά όργανα πολύ δρόμο. Έχουμε πολλούς νόμους, έχουν ληφθεί πολλές πολιτικές αποφάσεις μέσα ε, πρότυπα, στάνταρ και μη στάνταρ και έχουμε κάνει πολλά βήματα για να αποφύγουμε μια χειρότερη κρίση και να ξαναφέρουμε το τρένο που έχει εκτροχιαστεί στο σωστό δρόμο ε, για να παραμείνει σε αυτή την τροχιά και να ε, επανέλθει η εμπιστοσύνη. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας. Επανειλημμένα αναφερθήκαμε στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Ο κόσμος δεν έχει δει κανένα αποτέλεσμα που δεν θα μπορούσε άλλωστε ε, να το δει ακόμα. Και έχω την ερώτηση που είναι η εξής. Ε, θα κάνετε μια επισκόπηση ε, της ποιότητας των ενεργητικών και της υπόλοιπης ποιότητας των τραπεζών. Υπάρχει ένας κίνδυνος ε, να εμφανιστεί έτσι ένα πρόβλημα από καιρούς καιρών. Πώς εμείς θα αποφύγουμε με την πρώτη αρνητική είδηση να δημιουργηθεί πανικός. Πώς θα το αποφύγουμε αυτό, τον πανικό και το χάος. Το έχουμε υπόψη μας. Ξέρουμε ότι η εμπιστοσύνη δεν έχει ανακτηθεί επαρκώς για να είναι αρκετά σταθερή ε, σε κραδασμούς και στο παραμικρό αρνητικό νέο που θα προκύψει. Μεταξύ των θεσμικών οργάνων το συζητάτε αυτό. Έκανα την ίδια ερώτηση στον Επίτροπο Μπαρνιέ, ο οποίος μου είπε, το είπα στους Υπουργούς Οικονομικών και εγώ στο προηγούμενο ΕΚΟΦΗΝ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία και να ε, το έχουμε υπόψη μας και να μην εκπλαγούμε με την πρώτη αρνητική είδηση και την πρώτη δυσάρεστη. Αλλά πώς μπορούμε εκ των προτέρων να θωρακιστούμε καλύτερα. Ή μήπω ανησυχώ χωρίς ε, λόγο. Όχι, όχι. Ε, είναι πάρα πολύ εύστοχη η ανησυχία σας. Σε καμία περίπτωση δεν ανησυχείτε χωρίς λόγο. Και εμείς συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία και γνωρίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα και να είμαστε και προετοιμασμένοι. Η εμπειρία του παρελθόντος είναι πολύ κατατοπιστική. Τα πράγματα αυτή τη φορά είναι κάπως καλύτερα και γιατί οι τράπεζες έχουν αυξήσει σημαντικά τις προμήθειές τους και έχουν ε, ε, το κεφάλαιο τους αυξήσει σημαντικά. Η γενική κατάσταση και η εμπιστοσύνη είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα τεστ ε, κοπόσεως που έγιναν στις τράπεζες. Αλλά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα ε, χρειάζεται ε, επισκόπηση όλων των σημαντικών μηχανισμών και οργανισμών που θα ελέγξουμε. Είναι πολύ νωρίς από τώρα για να πούμε ε, ποιο ε, ποσό θα προκύψει, ποιο στοιχείο. Πιστεύουμε ότι αυτή η αξιολόγηση θα αυξήσει και τη διαφάνεια αλλά και την εμπιστοσύνη συνεπώς με την προϋπόθεση ότι ε, θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ε, κάποιες ελλείψεις. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή για τα εθνικά αποθεματικά και τα, εθνικά συστήματα που είναι απολύτως ε, απαραίτητα για να εξασφαλίσουν ε, την αξιοπιστία και των τεστ κοπόσεων και ε, των στοιχείων ενεργητικού. Αλλιώς θα υπάρξει παρερμηνία. Επειδή δεν υπάρχει καμία εθνική μέρεμνα, βγάζουν αυτά τα στοιχεία για να μην βγάλουν χειρότερα. Και τότε ε, αυτό πραγματικά θα ε, υπονομεύσει την αξιοπιστία του όλου εγχειρήματο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ε, με όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότητα, αλλά και συνέπεια παντού. Θα πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε σε περίπτωση που προκύψει κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα από τη, τους φιλελευθέρους ο Ραμόν Τριμόσα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Ντράγκη. Δύο ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Ε, ε, θα... Η Κεντρική Τράπεζα θα επιβλέψει κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες και χαίρομαι εγώ σαν Ισπανός που θα εποπτεύεται και των Ισπανικών τραπεζών. Το θέμα είναι όμως ποιος πρέπει να πληρώνει για τα λάθη της εποπτείας αυτής. Το δεύτερο θέμα που αφορά πάντα την εποπτεία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σωστή εποπτεία χωρίς αξιοπιστία. Η αξιοπιστία απαιτεί κάποιες τράπεζες να πτωχεύσουν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να έχει το κόκκινο κουμπί για να πιέσει για τη διάλυση μιας τράπεζας γιατί βλέπουμε σε ορισμένες χώρες, οι οποίες είναι πτώχευση σε ορισμένες χώρες, αυτό σημαίνει τεράστιες ε, ζημίες για τα κράτη-μέλη, για τους πολίτες τους, κοινωνικές περικοπές. Ξέρουμε τι έγινε στην Γερμανία με την West που πιέστηκαν έτσι ώστε να πτωχεύσουν. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για την πτώχευση ή μη μιας τράπεζας με λίγα λόγια. Για την πρώτη σας ερώτηση εγώ δεν θα ήθελα να σκεφτώ για το ποιος θα πρέπει να πληρώσει αν κάνει λάθος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά για το δεύτερο θέμα το οποίο θέσατε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Είπαμε εξ αρχής ότι η στιγμή κατά την οποία γίνεται η αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός πιστητικού ιδρύματος και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί πλέον το συγκεκριμένο αυτό πιστοτικό όργανο είναι δύο διαφορετικές στιγμές, δύο διαφορετικές εισαγωγικά αποστολές και πρέπει να γίνονται από δύο διαφορετικά όργανα. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι αυτή η οποία θα πει στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, το SRM, ότι ένα τάδε πιστοτικό ίδρυμα δεν είναι βιώσιμο. Και έτσι λοιπόν το SRM όπως και το FDIC στις Ηνωμένε Πολιτείε θα αποφασίζει το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο πιστοτικό. Αν θα πρέπει να πολιθεί, αν θα πρέπει να ανακεφαλαιωθεί, αν θα πρέπει να συγχωνευθεί ή αν θα πρέπει να πολιθεί εκ νέου και να διαλυθεί. Λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες οι οποίες κάθε φορά μπορεί να επηρεάζουν και τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα χρήματα των φορολογουμένων και ε, είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ανήκει στις αρμοδιότητες του SRM και είναι εντελώς διαφορετικές από τις αρμοδιότητες του επόπτη. Έτσι δουλεύει έτσι και αλλιώς και στις διάφορες χώρες μας. Έχετε τον επόπτη ο οποίος λέει στις υπεύθυνες αρχές, το Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι ε, ένα πιστοτικό ίδρυμα δεν είναι βιώσιμο και είτε πρέπει να στοχεύσει ή να συγχωνευτεί ή οτιδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει. Πάντως οι δύο αυτές αρμοδιότητες από ό,τι γνωρίζω σε όλες τις χώρες ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς κάθε φορά. Θέλετε να επανέλθετε σε αυτό. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία συζητάμε και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. how much flexibility την οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών. Οι διάφορες τράπεζες θα πρέπει ίσως να πτωχεύουν αλλά με διαφορετικό τρόπο όταν χρειάζεται. και οι, εξε, εξετάσεις από τις οποίες περνάνε κάθε φορά μπορεί να δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Μάριο, έχω μια ερώτηση για σένα σχετικά με τις μακροπροληπτικές ε, δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η μακροπροληπτική σας πολιτική είναι ένα σημαντικό νέο μέσο το οποίο μπορεί να ασκηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν αναλάβει το νέο της ρόλο στα πλαίσια του SSM, του ενιαίου μηχανισμού. Υπάρχει και μία πλευρά της μακροπροληπτικής η οποία αφορά και την προσπάθεια αντιμετώπισης ε, του συστήματος καθορισμού των επιτοκίων σε επίπεδο κρατών μελών δεν λειτουργούν σωστά και αυτό δημιουργεί πιέσεις για τα πιστοτικά ιδρύματα. Ποιος θα φροντίζει να ρυθμιστούν αυτές οι διαφοροποιήσεις και πώς ε, θα φροντίσετε έτσι ώστε η μακροπροληπτική πολιτική να εφαρμόζεται και σε επίπεδο εποπτείας αλλά και σε επίπεδο καθημερινής πολιτικής δηλαδή καθορισμού επιτοκίων κτλ. στην Τράπεζα της Αγγλίας ας πούμε, αυτό είναι μία από τις αρμοδιότητές τους. Κοιτάξτε, το εξετάζουμε ακόμα. Η μακροπροληπτική πολιτική, λέει ο πρόεδρος Ντράγκη, θα ενταχθεί και στα πλαίσια της εποπτικής αρχής και στα πλαίσια ε, του Συμβουλίου Διακυβέρνησης αν θέλετε. Εμείς προσπαθούμε να ορίσουμε σωστά τους τρόπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε μέσω έκτακτων συνεδριάσεων γύρω από τέτοιου είδους θέματα, έτσι ώστε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες κτλ. Δεν έχουμε καθορίσει ακόμα λοιπόν τις τελικές ρυθμίσεις. Να μην ξεχνάτε επίσης ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουμε και το θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Είναι λοιπόν αυτό που είπατε κάτι το οποίο μας απασχολεί και είναι κάτι το οποίο ακόμα ε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι αν θέλετε να ορίσουμε σωστά, να διευκρινίσουμε και προς εσάς έναν σωστό τρόπο, έναν έλογο τρόπο αντιμετώπισης του. Πρόκειται για ένα για έναν τομέα ο οποίος θα τον χαρακτήριζα φαιό, αδιαμόρφωτο ακόμα. Προσπαθούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την νομισματική πολιτική από τη μακροπροληπτική πολιτική και αυτό διευκολύνεται από τη συνθήκη. Ξέρετε ότι η βασική μας ευθύνη η σταθερότητα των τιμών μέσω πρόθεσμα, ξεκάθαρα. Αυτό κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη. Γιατί γνωρίζουμε ότι ανεξαρτήτως του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βασική μας εντολή είναι η διατήρηση των τιμών, η σταθερότητα των τιμών. Πέραν αυτού βέβαια μπορεί να υπάρχουν κάποια επιμέρους προβλήματα, τοπικά προβλήματα, σε έναν χώρο τόσο περίπλοκο όσο η Ευρωζώνη και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει εμείς να ασχολούμεθα με τοπικές φούσκες σαν παράδειγμα αν υπάρχουν ε, σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κάτι όμως το οποίο συνολικά επηρεάζει την νομισματική πολιτική. Η το κάνει αυτό ή μέσω του υποπτικού μηχανισμού. Ναι, ε, τώρα αυτές τις μέρες αυτό συζητάμε, τον καταμερισμό, ποιος θα κάνει τι. Α, μάλιστα. Δύσκολο αυτό το θέμα που σημειώσαμε. Έχουμε λίγο χρόνο και ε, ε ένα συνάδελφος που δεν ήταν εγγεγραμμένος για ερώτηση μου ζητάει το λόγο. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον Ιούλιο του 2012, κύριε Πρόεδρε, κάνετε μια ιστορική δήλωση, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να σώσει το ευρώ. Ε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια καθοδήγηση ε, πραγματικά σωστή προς τα εμπρός γιατί είχε σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στη νομισματική πολιτική περισσότερο στη δημοσιονομική ε, και έσωσε πολλές ε, χώρες από τη χρεοκοπία. Αλλά όπως έχει ήδη αναφερθεί ο μηχανισμός νομισματικής μεταβασής δεν είναι πραγματικά τέλειος γιατί είναι πολύ μικρή η ανάπτυξη των πιστώσεων και πολύ μικρή η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Δεν είναι η ηρωνία της ιστορίας αυτή ότι η δήλωση που κάνατε και τόσο φωτισμένη ε, τελικά ήταν υποστήριξη της δημοσιονομικής πολιτικής παρά ε, τόνωση της πραγματικής οικονομίας μέσω της νομισματικής πολιτικής. Συμφωνώ ότι το OMT ήταν πολύ αποτελεσματικό. Δεν συμφωνώ ότι ήταν ε, για ενίσχυση της δημοσιονομικής πολιτικής. Σε καμία περίπτωση το OMT είναι μια ε, μορφή και ένα εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εκείνη την εποχή οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζαμε μέσω του OMT ήταν κίνδυνη ε, ανα χαρακτηρισμού όπου είναι ένα εφημισμός ε, αυτός ε, και ουσιαστικά διεκβεβόταν η ίδια η ύπαρξη του ευρώ. Και ορισμένα από τα επιτόκια στην Ευρωζώνη δεν ε, το από τα βασικά στοιχεία της οικονομίας αλλά από αυτή την ε, αυτοπληρούμενη προφητεία ας πούμε ε, ότι θα διαλυόταν το ευρώ. Και αυτό ήρθε να κάνει εκείνη η παρέμβασή μας στην εποχή και ήταν στόχος νομισματικής πολιτικής γιατί υπήρχαν τέτοια καταστροφικά σενάρια τα οποία εμπόδιζαν ε, να φτάσουμε και να εκπληρώσουμε εμείς τη βασική μας συντολή που είναι η μεσοπρόθεσμη εγγύηση σταθερότητας των τιμών. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος. Γνωρίζετε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ε, να ε, πυροδοτείτε το OMT ε, στο μακροοικονομικό πρόγραμμα με τη δυνατότητα ενίσχυση από μια χώρα και αδυναμία προσφυγής αλλού. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου η πρόθεσή μας να αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα διαφόρων κρατών με την κίνηση αυτή. Ε, η υποκείμενη πεποίθησή μας είναι και ήταν και τότε και παραμένει ότι αν μια χώρα έχει μια δημοσιονομική θέση μη βιώσιμη, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα, κανένας άλλος για να την καταστήσει βιώσιμη, παρά μόνο η ίδια η χώρα. Και η βιωσιμότητα θα πρέπει να εκτιμάτε στους, ε, στα επιτόκια που αντανακλούν τα θεμέλια ε, ε, της οικονομίας και αυτό ήταν και στη βάση του σχεδιασμού της παρέμβασής μας μέσω των OMT. Άλλη μια ερώτηση θα δεχθούμε από τον Φιλίπ Λάμπερτς και μετά θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα που ζήτησε ο Μάριο πριν το επόμενο σκέλος ε, της ακρόασης για το συστημικό κίνδυνο. Η Σάρον ε, με κοίταξε προειδοποιητικά, θα είμαι σύντομος λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι οι χορηγήσεις προς την πραγματική οικονομία ε, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κλάδου των τραπεζών. Μα μήπως έχουν συνηθίσει αυτοί να έχουν απόδοση ε, που ε, δεν ε, συνάδει με την πραγματική οικονομία και μια σταθερή πραγματική οικονομία. Ναι, όντως. Όντως, για να απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, τι βλέπουμε σήμερα και τι παρατηρούμε. Όλοι οι κανονισμοί και η ρύθμιση ε, στους οποίους έχουμε προχωρήσει από τη χρηματοοικονομική κρίση και ε, μέχρι τούδε και συνεχίζουμε έχουν γίνει έτσι ώστε το τραπεζικό σύστημα και γενικά το χρηματοοικονομικό σύστημα να είναι λιγότερο ε, επικίνδυνο, δηλαδή να είναι μικρότερο το ρίσκο. Βεβαίως είναι σήμερα μικρότερη απόδοση σε σχέση με το παρελθόν γιατί ξέραμε ότι πραγματικά είχαν εθιστεί σε μία απόδοση που δεν είναι βιώσιμη στο δινεκές. Τώρα, με χαμηλότερη απόδοση, αυτό σημαίνει σήμερα ότι είναι και χαμηλότερος ο κίνδυνος. Αυτό χρειάζεται χρόνο για να εδρεωθεί και να συνηθίσουν οι αγορές, ε, οι τράπεζες, να το εκτιμήσουν και να το εμπεδώσουν. Ότι η απόδοση θα είναι χαμηλότερη, αλλά θα παραμείνει και χαμηλότερη. Ταυτόχρονα μειώνεται και το ρίσκο και ο κίνδυνος. Άρα είναι διαφορετικός ο συσχετισμός ρίσκου και απόδοσης και θα πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να συνηθίσει σε αυτό. Βέβαια η σημερινή κατάσταση είναι κατά πολύ καλύτερη από ό,τι πριν από μια τριετία. Όπως βλέπετε οι τράπεζες και πάλι μπορούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια, να δανείζονται από τις αγορές. Ε, έχει βελτιωθεί γενικά η κατάσταση από πλευράς εμπιστοσύνης. Ε, σιγά σιγά ε, καταλαβαίνουν οι ενεχόμενοι το νέο περιβάλλον. Ότι είναι μεν χαμηλότερη απόδοση, αλλά είναι χαμηλότερο και το ρίσκο και αντίστοιχα συμπεριφέρονται και ανταποκρίνονται. Όπως σας είπα προηγουμένως για την επισκόπηση της ποιότητας του ενεργητικού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλέον διότι για να πείσει κανείς τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στις τράπεζες, τι χρειάζεται. Όχι μόνο χαμηλότερο κίνδυνο, αλλά και διαφάνεια ε, στους ισολογισμούς των τραπεζών. Γι' αυτό μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι ε, ροές ε, ε, από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία. Thank you very much. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Φτάνουμε και στο τέλος της, του σκέλους νομισματική πολιτική. Όπως σας είπα θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, πεντάλεπτη, και θα αρχίσουμε με την επόμενη ακρόαση λίγα λεπτά νωρίτερα, αλλά έτσι επιτρέπουμε και στο Μάριο να φύγει ενδεχομένως λίγο νωρίτερα. Σε πέντε λεπτά επιστρέφουμε. Right. Καλώς ήρθατε και πάλι συνάδελφοι. Θα περάσουμε τώρα στην ακρόαση πάλι με τον πρόεδρο αλλά με διαφορετική ιδιότητα. Την ιδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Θα κάνει λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις με αυτή του την ιδιότητα και θα περάσουμε στις ερωταπαντήσεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Μάρια, ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι ενώπιον τη Επιτροπή σα σήμερα για να σε ενημερώσω για τι δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα πω ότι στην περασμένη συνεδρίαση ο διοικητή Κάρνη τη Τράπεζα τη Αγγλία διορίστηκε αντιπρόεδρο, πρώτο αντιπρόεδρο τη ΕΚΤ. Ε, από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε είδαμε ενδείξεις αλλαγής των οικονομικών προοπτικών της Ευρώπης, σταδιακής αλλαγής. Είναι ενθαρρυντικές οι εξελίξεις και όπως πολλές φορές σας είπα βρίσκονται στην παιδική του ηλικία αυτές οι αλλαγές. Παρόλα αυτά ελοχεύει ο κίνδυνος σε σχέση με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα ήθελα να σας πω με ποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου κινείται για να καλύψει αυτούς τους κινδύνους στους τομείς των ασφαλιών, τον τραπεζικό τομέα και ως προς τις υποδομές της αγοράς. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω σε σχέση με δύο τομείς αξιολόγηση της εφαρμογής της πρώτης σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση μακροπροληπτικών εργαλείων προσαρρογή των εθνικών αρχών. Ε, ο τομέας των ασφαλιών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ευρύτερα στην οικονομία. Πέρα από την ανάληψη κινδύνων που τα νοικοκυριά ή οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να υπομισθούν ε, τα ίδια, λειτουργεί και ως επενδυτής ο τομέας των ασφαλείων. Ε, ταυτόχρονα ε, υφίσταται η ανάγκη αντιμετώπισης ε, των πιθανών κινδύνων και ευπαθών καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν για τις ασφάλειες και μπορεί να επηρεάσουν γενικότερα τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες για ασφάλειες ζωής, κυρίως όσες έχουν εγγυημένες αποδόσεις, πλήττονται λόγω του περιβάλλοντος των χαμηλών υψηλών επιτοκίων. Εάν τώρα το εξετάσουμε αυτό το δεδομένο από μικροπροληπτική σκοπιά, ο ΕΙΟΠΑ συνέστησε σωστά στις επιχειρήσεις να τροποποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Αυτό έχει κέρια σημασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην οικονομική του πηγή. Εάν τα επιχειρηματικά μοντέλα δεν τροποποιηθούν, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίζουν να επιδιώκουν υψηλότερες αποδόσεις, επενδύοντας σε πιο επικίνδυνα χρεόγραφα. Όμως αυτό ε, συνεπάγεται ενδεχομένως ε, ε, μεγάλες απώλειες λόγω των αυξήσεων στα ασφάλιστρα. Έχουν περιορίσει τα κίνητρα οι ίδιες επιχειρήσεις εάν τα κανονιστικά καθεστώτα δεν τονίσουν αυτούς τους κινδύνους. Ο τομέας έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει την οικονομία και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε ποιες παρά παράπλευρες επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν για το γενικότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω άμεσων συνδέσμων με την πραγματική οικονομία και κοινών σημείων έκθεσης. Ε, είναι συστημική σημασία λοιπόν ο τομέας των ασφαλιών ε, και αυτό το συνειδητοποιούμε όλο ένα και περισσότερο. Το ε, Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εσχάτως ανακοίνωσε ένα κατάλογο συστημικώς σημαντικών παγκοσμίων ασφαλιστικών ομήλων, πέντε εκ των οποίων είναι ευρωπαϊκοί. Η Διεθνής Ένωση των Ασφαλιστικών Εποπτών έχει αναπτύξει πλαίσιο για απόκριση από πλευρά πολιτικής ε, συμπεριλαμβάνοντας και μια δυνατότητα, αυξημένη δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών και αποτελεσματικής λύσης και καθάρισης οργανισμών. Στη ΣΥΠΑ οι συστημικά ε, σημαντικές ε, συστημικά σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί όπου συμπεριλαμβάνονται και ασφαλιστικές εταιρείες θα υφίστανται εποπτεία από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΦΕΔ. Στην Ευρώπη ε, το νέο σύστημα προληπτικής ε, ρύθμισης ε, φερεγγιότητα 2 συνεχίζεται και από αυτή την πλευρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει κέριο ρόλο διότι είναι συνομοθέτης. Η φερεγγιότητα 2 απηχεί το προφίλ ρίσκου των ασφαλιστικών εταιριών πολύ καλύτερα σε σχέση με τη φερεγγιότητα 1 και ενισχύει την ικανότητά τους για τη διαχείριση κινδύνων. Ταυτόχρονα το νέο σύστημα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις πιθανές και ε, μίες και μένες επιπτώσεις αυτής της ε, βραχυπρόθεσμης πτυτικότητας των αγορών ε, ε, καλύπτοντας και τις προκυκλικές επιπτώσεις όπως τα LTROs κάνουν αυτή τη στιγμή και όλα τα πακέτα που εγγυήσεων. Όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ESRB έχει συμμετάσχει στην οικονομική αξιολόγηση του πακέτου εγγυήσεων που διεξάγει ο ΕΙΟΠΑ και υποστηρίζει τα βασικά συμπεράσματα. Δεδομένου όλων αυτών των στοιχείων που προανέφερα είναι κέρια σημασία στο πακέτο αυτό να καλύψει και επαρκή επίπεδα κεφαλαιακά αλλά ταυτόχρονα και ε, αδιάκοπα ε, πλήρη διαφάνεια ως προς την εφαρμογή. Ε, θα έπρεπε λοιπόν κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους που ελοχεύουν. Τώρα το τραπεζικό σύστημα επίσης έχει κέριο ρόλο να παίξει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ταυτόχρονα ο ρόλος κατά την εκδίπλωση της χρηματοπιστωτικής κρίση, κρίσης τόνισε ε, και το πω στη, την ευπαθή θέση στην οποία βρίσκεται. Χρειάζονται σημαντικά βήματα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και ούτως ώστε να έχουμε ένα υγιέστερο τραπεζικό σύστημα που αξίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, και αυτό είναι ένας τομέας ε, όπου το το Κοινοβούλιο έχει παίξει καταλητικό ρόλο εγκρίνοντας τον κανονισμό για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό των SSM. Η επερχόμενη συνολική τραπεζική αξιολόγηση που διεξάγει η ΕΚΤ, που διεξάγεται με τρόπο ε, που συμμορφώνεται πλήρως με τις ε, συνστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπως εξαγγέλθαν το Μάρτιο του 2013, έχει την δυνατότητα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε σχέση με την υγεία ε, και την, το αν την αποτελεσματικότητα του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Αυτό θα μείωνε το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών, άρα και της χορήγησης πίστης για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Αυτό χρειάζεται πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική. Επίσης, εξάντε χρειάζονται με αξιόπιστοι αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου, καθώς και δημοσιονομικά αποθέματα, ε, αν παραστεί η ανάγκη, για να απορροφηθούν κεφαλαιακές ελλείψεις που θα εντοπιστούν από μια ε, μελλοντική αναθεώρηση. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου εξετάζουμε δύο διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματο ε, που ε, ήρθαν στο φω με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Πρώτον, το μεγάλο μέγεθο του τραπεζικού συστήματο ε, σε σχέση με το μέγεθο πραγματική οικονομία και δεύτερον, η συγκέντρωση των απολειών σε ορισμένου τομεί τη χορήγηση πίστη. Σε πολλέ χώρε βλέπουμε ότι αυξάνονται με οργού ρυθμού τα ενεργητικά των τραπεζών και η μόχλευση το ίδιο. Αυτό δεν είναι βιώσιμο βιώσιμο. Μόλις ε, προκύπτουν ε, πιστοτικές απώλειες, ε, είδαμε ότι οι χώρες χρειάστηκε να στηρίξουν τον τραπεζικό τομέα υποπίεση και επιδίωξαν απομόχλευση, περιορίζοντας έτσι και την προσφορά πίστη στην πραγματική οικονομία. Αυτό διεύρυνε την κρίση εντείνοντας την ύφεση και εμποδίζοντας την ανάκαμψη. Με αυτό υπόβαθρο το Γενικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου εξακολουθεί να εξετάζει το Πώ το μέγεθος του τραπεζικού τομέα σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας επηρεάζει ε, την προσφορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εποφελών από κοινωνικής πλευράς. Ε, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου άρχισε να πραγματεύεται ακριβώς αυτό το ζήτημα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι απώλειες των τραπεζών συγκεντρώθηκαν όπως σας έλεγα σε ορισμένους τομείς της δανειοδοσίας. Σε ένα ορισμένο αριθμό χωρών οι απώλειες σε σχέση με τα ενυπόθηκα δάνεια παραδείγματος χάρη κατέστησαν ήταν αναγκαίες παρεμβάσεις δημόσιες μεγάλης κλίμακας στον τραπεζικό ε, τομέα, αλλά ακόμη και τομείς νης ε, εξειδικευμένοι όπως η ναυτιλία παραδείγματος χάρη, ε, χρειάστηκαν παρέμβαση σε μεμονωμένες τράπεζες σε κάποιες χώρες. Κυκλικοί τομείς όπου έχουν μεγάλη έκθεση οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο κατασκευαστικός τομέας και τα κτηματομεσητικά, καταναλωτικά πάγια αγαθά όπως παραδείγματος χάρη η αυτοκινητοβιομηχανία, υλικά και ε, προϊόντα μεταποίησης, ε, χαλιβουργία και χημική βιομηχανία ε, παρουσιάζουν τις ίδιες τάσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν στις εργασίες μας σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο ρόλο των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Είναι στοιχείο κλειδί στην χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι οι χώρες G20 έχουν συμφωνήσει ότι όλες οι τυποποιη... όλα τα τυποποιημένα παράγωγα, τα έξω χρηματιστηριακά κατά τα over the counter πρέπει να εκαθαρίζονται από, τέτοιους, από τέτοια αντισυμβαλόμενα μέρη και τα αντισυμβαλόμενα μέρη όντως έχουν το όφελος της μείωσης του κινδύνου αλλά ταυτόχρονα έχουν συστημική σημασία διότι είναι ε, κέρι βρόχη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό συνεπάγεται μακροπροληπτικούς κινδύνους. Η κυκλικότητα ε, των κανόνων περιθωρίου των αντισυμβαλλωμένων ε, μερών και οι πρακτικές τους είναι βασική μας ανησυχία. Το να αυξηθούν τα περιθώρια σε περιπτώσεις ε, κρίσης και μείωση σε περιπτώσεις οικονομικής ευημερίας μπορεί να έχουν νόημα όταν εξετάζει κανείς το θέμα από τη σκοπιά ενός αντισυμβαλλωμένου μερός. Όμως ελοχεύει ο εξής κίνδυνος να αυξηθεί η κυκλική ευπάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος η οποία μπορεί να αυξηθεί στο μέτρο της που έχει το κάθε συμβαλόμενο μέρο Και ο ΕΣΜΑ παρότι έχει εντάξει ε, κάποιες σε διατάξει μέσα στα τεχνικά της ε, πρότυπα, η αποτελεσματικότητά του από μακροπροληπτική πλευρά ε, μπορεί να ενισχυθεί από άλλα μέτρα μετριασμού αντικυκλικού όμω χαρακτήρα. Τα αντισυμβαλόμενα μέρα επίσης χρειάζονται κρατεά σχέδια ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών για να αποφύγουμε μια άτακτη χρεοκοπία και αφαιρεγγιότητα. Τέλος, ε, υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης ε, κυρίως ε, στα συμβαλόμενα μέρη που εκαθαρίζουν τα ίδια προϊόντα βάσει των επωνομαζόμενων ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας. Οι αναπτυσσόμενες αγορές αντισυμβαλωμένων μερών πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε να μειώνουν τις παράπλευρες απώλειες μιας ενός ενδεχόμενου προβλήματος από τον έναν αντισυμβαλόμενο στον άλλον. Και γι' αυτό το στόχο ο ΕΣΜΑ έχει ήδη εκδώσει ειδικέ κατευθυντρίε γραμμέ. Ε, παρόλα αυτά, δεδομένε τη συστημική σημασία των αντισυμβαλωμένων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ευρύ οπλοστάσιο εργαλείων για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά ω προ την επιμόλυνση. Η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει στο Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έναν πολύ ξεκάθαρο ρόλο σε αυτού του τομεί. Παραδείγματο χάρη βάσει των διατάξεων ε, του ΕΜΙΡ, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού δηλαδή για την υποδομή των αγορών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, καλείται να εξετάσει τις επιπτώσεις της προκυκλικότητας των πρακτικών περιπεριθωριών των αντισυμβαλωμένων μερών και να εποπτεύσει το σχεδιασμό των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Στιμικού Κινδυνού θεωρεί, ε, εξετάσει μάλλον αυτά τα ζητήματα στην τελευταία διάσκεψη που είχε σε επίπεδο Γενικού Συμβουλίου και έχει σχεδιάσει τη μελλοντική δική της ε, εργασία γι' αυτό. Τώρα, τι έπεται. Μελλοντικέ εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα εφαρμογή τη πρώτη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κίνδυνου. Όπω ξέρετε, οι συστάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι εργαλεία soft όπω ονομάζονται, όχι νομοθετικού χαρακτήρα δηλαδή και συνοδεύονται από ένα μηχανισμό actor explain. Δράστη εξηγήστε γιατί όχι. Έτσι, από πλευρά λογοδοσία είναι σημαντικό να αξιολογούνται οι δράσει των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων εξηγήσεων για έλλειψη δράση με το που εκδοθεί μια σύσταση του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου στημικού Κινδύνου. Για την πρώτη του λοιπόν σύσταση για τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις ολοκλήρωσε τον πρώτο ε, πλήρη κύκλο από την έκδοση δηλαδή της σύστασης έως και την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής. Όπως θα θυμάστε ίσως, η σύσταση θεσπίζει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών συστημικών κινδύνων κατά το δανεισμό σε ξένο νόμισμα προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα. Το Γενικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την αξιολόγηση που θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες και ο στόχος είναι να εφαρμοστεί παρεμφερή σε διαδικασία και για τις επόμενες αξιολογήσεις των άλλων συστάσεων του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με την καθοδήγηση για τη χρήση των μακροπροληπτικών εργαλείων που ε, προβλέπεται στους ε, πρόσφατα εγκεκριμένους ευρωπαϊκούς ε, και κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια. Ξέρετε ότι θα αρχίσουν να ισχύουν σχετικοί κανόνε το 2014 και προβλέπουν ένα φάσμα μακροπροληπτικών εργαλείων που οι εθνικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους προς χρήση. Όπως σας είπα και στην προηγούμενη ακρόαση στις 8 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο Στιμικού Κινδύνου συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για τις καθοδηγήσεις που θα δώσει ως προς τον τρόπο χρήσης από πλευρά των εθνικών αρχών αυτών των εργαλείων με συντονισμένο τρόπο και θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη ακρόαση για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε και για το διορισμό του πρώτου αντιπροέδρου. Ήδη διερευνούμε εάν μπορούμε και πότε μπορούμε να κάνουμε ε, μια ακρόαση, μάλλον αρχές του επομένου έτους, γιατί ε, είναι μεγάλος ο φόρτος εργασίας, πάντως θα γίνει. Όπως είπατε, και αναφερθήκατε στις ασφάλειες και έχουμε εργαστεί πολλοί από εμά αρκετά σκληρά για να ολοκληρωθεί η φερικιότητα 2 εντός του πλαισίου του οδηγίας ε, και των προτάσεων Omnibus 2. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες, αλλά ε, στα συστημικά πλαίσια οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, είναι όλο και πιο συστημικές γιατί τώρα απειλούνται με bail-in και ένα σύστημα εξυγίασης τραπεζών. Ενώ στο παρελθόν ε, έμεσα και σιωπηρά υπήρχε εγκύρηση των τραπεζών. Δηλαδή είναι μια νέα ατζέντα συστημικού κινδύνου αυτή και θα τις περιλαμβάνει. Η έννοια ε, του τι είναι συστημικό διαφέρει από τις τράπεζες, τις ε, ασφαλιστικές εταιρείες τράπεζα έχει να κάνει με το bank run και ενδεχομένως ε, τα προβλήματα ρευστότητας να γίνονται προβλήματα φερεγγιότητας. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες τι σημαίνει να είναι συστημικές. Ε, ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες όπως η διαφοροποίηση του κινδύνου ε, χάνονται. Ας πούμε δεν θα υπάρχει αντασφάλιση. Επίσης μακροπρόθεσμα όταν ε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση ε, της οικονομίας ή όταν προκυκλικά θα πρέπει εκτάκτως να πολλούν μαζικά. Ε, fire sales. Και επίσης οι διάφοροι μηχανισμοί που έχουν δημιουργηθεί για τη μακροπροληπτική εποπτεία έχουν εντοπίσει στο FSB και IIS πέντε από εννέα ασφαλιστικές εταιρείες ε, είναι ευρωπαϊκές σας είπα, ε, παγκοσμίως συστημικές δηλαδή. Άρα υπάρχει διαφορετική εκτίμηση για το τι είναι συστημικό. Ε, αν πρόκειται για τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία. Δεν είναι μόνο το bail-in, αλλά υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Να σας πείσω λίγο παραπάνω από μια άλλη σκοπιά. Ε, αναφερθήκατε στη μακροχρόνια επένδυση. Τώρα γίνονται διάφορες ε, προτάσεις να προσπαθήσουμε ε, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιωτικά ταμεία να ενδιαφέρονται περισσότερο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αλλά ζητούν κάποια εγγύηση για αυτές, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από κάπου αλλού. Αν βάλετε λοιπόν κάπου κυβερνητικές κρατικές εγγύησεις στη μακροπρόθεσμη επένδυση από πλευράς ασφαλιστικών εταιριών τελικά μήπως μεταφέρεται από την τράπεζα τι επιδοτήσει των τραπεζών για μακροπρόθεσμε επενδύσει ουσιαστικά σε επιδοτήσει των ασφαλιστικών εταιριών για να κάνουν μακροπρόθεσμε επενδύσει. Ναι, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αυτός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών υπάρχει, ε, υπήρχε ανέκαθεν και υπάρχει θετική πλευρά σε αυτό, διότι έχουν ένα αντικυκλικό ρόλο. Οπότε αυτοί είναι οι βασικοί θεσμικοί επενδυτές ε, που έχουν κύριο ρόλο για τη χρηματοδότηση ε, κέριων υποδομών και επίσης παίζουν και ένα ρόλο κατά των βραχυπρόθεσμων κινήσεων που γίνονται στο οικονομικό σύστημα και ακόμη και χωρίς εγγυήσεις θα έλεγα ότι εσχάτως υπάρχει μια τάση μεγάλες ασφαλιστικές να μπαίνουν σε βραχυμεσοπρόθεσμα δάνεια για την χρηματοδότηση και λόγω της παγκόσμιας έλλειψης πίστης ε, καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει, υπάρχει υπαρκή ικανότητα διαχείρισης ε, των κινδύνων και διαχείριση των πιστοτικών κινδύνων. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζονται επιπρόσθετες ε, εγγύσεις, διότι ανέκαθεν είχε αυτή την επενδυτική πολιτική εκεί. Ωραία. Ε, ε μπορεί να ζητάνε ό,τι θέλουν, αλλά μπορεί να μην τους το δώσουμε εμείς. Λοιπόν, Διόγκο Φέιο, ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Σάρων, Πρόεδρε Ντράγκη, θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω και να σας πω ότι Μα, μ' άρεσε πάρα πολύ η αναφορά που κάνατε στη σημασία που έχει ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στις ε, οικονομίες των κρατών μελών της ευρωπαϊκή Ένωσης. Τι έχει σημασία σε αυτό το τομέα. Η εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι καταθέτες στο σύστημα και αυτό σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση. Ήδη και δικαίω έχουμε ε, ε, ε, εργαστεί επισταμένα για το ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με την εξυγίανση, τη λύση και καθάριση τραπεζών και την εγγύηση των καταθέσεων. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μόλις έμαθαν ότι υπάρχει η αρχή του bail-in και τελικά ε, ε, στο κάτω-κάτω στην ιεραρχία υπάρχουν καταθέσεις 100.000 ευρώ, ήρθαν σε επαφή μαζί μου με αυτήν την ε, ανησυχία και εγώ φυσικά αποκρίθηκα καθησυχάζοντάς τους. Όμως, Πρόεδρε Ντράγκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Στις μελλοντικέ μας εργασίες πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις χάρη στις οποίες θα έχουμε μια επιπρόσθετη εμπιστοσύνη για τους Ευρωπαϊκούς Ευρωπαίους καταθέτες. Απάντηση. Σε, ένα, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η καλύτερη υποστήριξη προς τους καταθέτες είναι ακριβώς η επιστροφή της εμπιστοσύνης ε, γενικότερα στο οικονομικό σύστημα και η παγίωση μιας ισχυρής ανάκαμψης. Ε, τώρα, ε, για το συγκεκριμένο θέμα της εξυγένσης των τραπεζών, ας κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους ομίλους που έχουν πια κλείσει και αυτούς που ακόμη λειτουργούν. Ε, για την πρώτη κατηγορία, όταν έχουμε το pecking order, δηλαδή την ε, ιεραρχία αυτών που θα αποζημιωθούν, ε, βλέπουμε ορισμένες φορές ότι υπάρχει αφενός προτίμηση για τους καταθέτες και αφετέρου bail-in για ε, τα χρεόγραφα. Ανάμεσα σε αυτούς θα έχουμε διάφορες κατηγορίες πιστωτών και έχουμε τώρα και τη δεύτερη κατηγορία των ομήλων, που βρίσκονται ε, σε προβληματική κατάσταση, εκεί πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα σε σχέση με το bail-in, στο μέτρο που εξακολουθεί να είναι βιώσιμη η τράπεζα. Η καλύτερη λύση που μπορούμε να δώσουμε, εν τη αυτή περίπτωση, είναι να έχουμε ένα σετ εργαλείων που θα έχουν αποφασίσει οι όμιλοι εκ των προτέρων και θα χρησιμοποιηθούν αν συμπληρούνται οι προϋποθέσεις για bail Και γι' αυτό είναι σημαντικός ο υποπτικός ρόλος ε, από αυτή την πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να επανέλθετε στην ερώτησή σας. Ναι, ήθελα να σας ζητήσω ένα σχόλιο για κάτι που έμαθα πρόσφατα. Ε, υπάρχει στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα μια επιχείρηση στην Πορτογαλία που τον Νοέμβριο του 2012 πλήρωνε ε, επιτόκιο 6,2 για ένα δάνειο. Σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι τρεις φορές μικρότερα τα επιτόκια. Πώς, πώς θα υπερβείτε αυτή την ανισορροπία που υπάρχει. Um, Η κατάσταση αυτή είναι προϊόν της οικονομικής κρίσης που δημιούργησε αυτή την πολυδιάσπαση στον χώρο της ζώνης ευρώ. Σε σχέση με το κόστος της χρηματοδότησης είδαμε ότι υπάρχουν βελτιωμένα στοιχεία για τις τράπεζες. Από την άλλη σε επίπεδο δανειστών είναι τα πράγματα λιγότερο καλά. Βλέπουμε ότι το κόστος της ε, δανειοδότησης ποικίλει φυσικά από χώρα σε χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει βέβαια και με το ότι δεν μπορούμε παρά να δεχθούμε ότι ο κίνδυνος ε, των δανείων στις πιεσμένες οικονομίες ε, είναι υψηλότερο από ότι στις χώρες που δεν αντιμετωπίζουν αυτό το λεγόμενο στρες. Στις πιεσμένες οικονομίες πολλές τράπεζες αγοράζουν σημαντικά τμήματα του χρέους του δημοσιονομικού τους. Και φυσικά το κόστος αυτό είναι ψηλότερο και η απόδοση από τις συγκεκριμένε αντίστοιχες ενέργειες τις οποίες προβαίνουν στις χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται σε πίεση. Αυτό δείχνει ίσως και το πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Η θα έλεγα σταθεροποίηση των ρυθμών ανάπτυξης, η σταθεροποίηση των μεταρρυθμίσεων. Θα αυξήσει την εμπιστοσύνη, θα μειώσει τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων και θα βελτιώσει την δανειοδότηση και την δανειοληψία επίσης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μερικές φορές η εξαγορά των ομολόγων είναι αυτή η οποία στεγνώνει την αγορά από δάνεια. Κοιτάξτε, είναι μια εναλλακτική μορφή επενδύσεων. Αν πράγματι τα επιτόκια ήταν χαμηλότερα, τότε οι τράπεζες θα δάνειζαν περισσότερο αλλά και με χαμηλότερο κόστος. Θα πρέπει να δει κανεί και την αποστροφή στους κινδύνους των πιστοτικών ιδρυμάτων στη σημερινή οικονομία να προσπαθήσει να δει κανεί ποια είναι η απόδοση σε σχέση με τον κίνδυνο. Αν η ανάκαμψη ήταν πιο ισχυρή, πιο εγκατεστημένη σε εισαγωγικά, τότε τα επιτόκια θα κατέβαιναν. Αν οι δημοσιονομικές προσπάθειες μεταρρύθμισης ήταν ισχυρότερες, τότε το κόστος θα ήταν χαμηλότερο και αν ήταν υψηλότερος και ο κίνδυνος επίσης ε, ε, και στα κρατικά ομόλογα και για τα πιστοτικά ιδρύματα τα οποία εκτίθενται σε αυτά, αυτό θα βελτίωνε τη δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Uh, Αυτή η ερώτηση είναι περίπλοκη, είναι δύσκολη. Από τη μία θα έλεγε κανείς ότι το να δανείζει κανείς τις κυβερνήσεις πιο ακριβά θα καταστήσει το να δανείζει τις επιχειρήσεις φτηνότερο, είναι με ένας ισχυρισμός. Από την άλλη, αν αυξήσει την απορροφητικότητα κεφαλαίων των κυβερνήσεων μέσω των κρατικών ομολόγων θα υπάρχουν λιγότερα κεφάλαια διαθέσιμα για την πραγματική οικονομία. Δεν είναι εύκολη λοιπόν η απάντηση πόσο θα επηρεάσει την αγορά η κατάσταση αυτή. Πέραν αυτού, αν θέλετε να σταθμίσετε τους κινδύνους με διαφορετικό τρόπο για τα δάνεια προς τις κυβερνήσεις, τότε οι κίνδυνοι αυτοί θα είναι πολύ ψηλότεροι φυσικά για τις πιεσμένες χώρες από ότι για τις μη πιεσμένες χώρες. Οπότε η απορροφητικότητα των κεφαλαίων θα είναι υψηλότερη για τις πιεσμένες χώρες από τις χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν το αντίστοιχο πρόβλημα. Βλέπετε ότι η απάντηση στην ερώτησή σας δυστυχώς είναι πολύ περίπλοκη. Γενικά έχουμε μπλέξει λέει πρόεδρος και δύσκολα θα βγούμε από αυτό το μπλέξιμο. Καντραουή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για την εισαγωγή σας. Εγώ θα μιλήσω ε, για την παρατραπεζική, της παρατράπεζες. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβαίνει σε μια ρύθμιση ε, για τα ταμεία που ε, χρηματοδοτούν τις τράπεζες βραχυπρόθεσμα αλλά και τα κράτη και ενδεχομένως έχουν και ένα συστημικό κίνδυνο. Η σταθερότητα ρευστότητας και εγγύησης αυτών των ταμείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση ακριβώς για να καλύπτει ενδεχόμενο συστημικό κίνδυνο πέραν και του κινδύνου υπερβολικής εμπιστοσύνης σε εξωτερική βαθμολογία που επηρέασε και στο παρελθόν, ε, γίνεται λόγος και ένα μεγάλο κίνδυνο ε, των λεγόμενων ε, runs που υπάρχουν έτσι πιο μεταβλητές βαθμολογίες. Υπάρχει μια οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσει ε, CNF 3% ε, προτείνεται. Νομίζετε ότι είναι καλή αυτή η προσέγγιση ή ε, κάτι άλλο που προτείνουν και άλλα κείμενά σας. Αυτά τα CNAF να απαγορεύονται και να περνάμε στα περίφημα VNAFs. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία της χρηματαγοράς ε, και τέτοια ταμεία που ε, πρέπει να καλυφθούν από πλευράς συστημικού κινδύνου. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δημόσια σύστασή μας του Δεκεμβρίου του 2012 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ταμεία ε, τα λεγόμενα money market funds και άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες όπως και στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν αντίστοιχες συστάσεις και μάλιστα εκεί αυτός ο κλάδος είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στην Ευρώπη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή ε, την ε, ιδέα, τα σύναυς που ε, είναι τα μία που έχουν σταθερή αξία στην αγορά, είναι αντίστοιχα περίπου με πιστό ερευνητικά ιδρύματα. Είναι περίπου αντίστοιχα με συστημικές τράπεζες και θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία ε, ε, έτσι ώστε να μεταβληθούν σε ε, στοιχεία μεταβλητής αξίας, βίναυς και όχι σύναυς. Υπάρχει μια περίπτωση φυγής εμπεδιτών, αλλά δεν είναι πάντα η δυνατότητα να επεμβαίνουν οι ρυθμιστές με τον ίδιο τρόπο που επεμβαίνουν στις τράπεζες. Στις 4 Σεπτεμβρίου ε, κατατέθη μία πρόταση κανονισμού ε, ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταθέτει μια διαφορετική πρόταση. Να μην απαγορεύονται τα σύναψ, αλλά να υπάρχει ακριβώς ένα buffer 3% ρευστού στα στοιχεία ενεργητικού και όταν δεν ε, είναι σε θέση τα ιδρύματα αυτά να ε, τηρούν αυτό το όριο, αυτόματα θα ε, καθίστανται βίνας. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις συστάσεις στις δικές μας είναι κάτι που θα μας απασχολήσει το 2014. Η απάντηση στην ειδική σας ερώτηση για το αν αρκεί το 3% ή όχι θα σας δοθεί εν ευθέτω χρόνο. Αυτή τη στιγμή Νομίζω υπάρχει αρκετά για να γνωρίζετε περίπου πού κινούμεθα. Ναι. Μήπως λίγο πιο γρήγορα να μας απαντήσετε και όχι το 14. Γιατί εμείς θα το κοιτάξουμε αυτό το θέμα πριν τα τέλη του έτους. Όλοι Σμιτ από τους φιλελευθέρους. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας χαιρετώ χαιρετίζω και σας συγχαίρω για τη νέα πολιτική για τα φύλλα στην ΕΚΤ, την ισότητα των δύο φύλων. Ε, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ακούσατε ε, τι λέει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο πάλι όχι. Έτσι ήταν κύριε Λάγκε, να αφήσετε τα αυτά. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, Πρόεδρε, τώρα την ε, για την οικοδόμηση της πραγματικής τραπεζι... ουσιαστικής τραπεζικής ένωσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο, στο πω έτσι, δεν ενδέχεται να είναι περίπλοκο και άρα ε, να δυσχεράνει την ανάληψη ε, ταχείας δράσης. Εγώ ε, είμαι από χώρα που είναι εκτός Ευρωζώνης, εγώ λυπούμαι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τι θα γίνει με τις τράπεζες εκτός Ευρωζώνης που έχουν θυγατρικές εντός, ε, καταστήματα εντός. Ε, και όταν είναι συστημικά σημαντικές και άρα επικίνδυνες, ε, τι θα γίνει, δεν θα κατονομάσω συγκεκριμένες ε, τράπεζες. Και μπορείτε να απαντάτε πραγματικά χωρίς να πείτε ούτε λέξη για τις χθεσινές εκλογές, μα είναι πολιτικό το όργανο και πολιτική αποστολή μας. αν κοιτάξω τι συμβαίνει στην αγορά αυτή τη στιγμή, είναι λίγο πτητική με, τις, ε, με το αποτέλεσμα των εκλογών τι θα γίνει, θα έχουμε μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη. Απάντηση. Θα ζητήσω να με εξαιρέσει η Πρόεδρος από απάντηση σε αυτό το ερώτημα και ελπίζω να γίνει δεκτό το έτοιμά μου. Για το πρώτο που ρωτήσατε, πώς μπορούν να συνεπάρχουν ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και ε, ε, με το ESSM με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Ε, μα είναι νέος θεσμός το e SSM, ενώ το ESRB έχει soft αρμοδιότητες, δεν είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις του όπως αυτές του e SSM. Ε, το e SSM ασχολείται μόνο με την Ευρωζώνη, ενώ το ESRB όχι. Το ESSM ε, θα αναλάβει κάποιες από τις λειτουργίες ε, που επιτελούν τώρα μέλη της ΕΚΤΕ, παραδείγματος χάρη για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα και θα έχει κοινέ αρμοδιότητες με τις εθνικές ε, μακροπροληπτικές αρχές στον τραπεζικό τομέα. Τα καθήκοντα του ESRB από το, για το CRR θα παραμείνουν στο ESRB επικάλυψη μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Συμβούλιο του ESRB. Γιατί πρέπει να έχουμε τακτική ροή πληροφοριών για τα μακροπροληπτικά εργαλεία. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει ικανοποιητική ε, ροή πληροφοριών. Η Επιστημονική Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε και μια σχετική μελέτη και σας παραπέμπω σε αυτήν διότι είναι ε, ενδιαφέρουσα τεκμηρίωση. Μετά με ρωτήσατε για τις τράπεζες ε, που δεν έχουν την έδρα τους στην Ευρωζώνη, έχουν όμως καταστήματα στην Ευρωζώνη, υποκαταστήματα. Τι θα γίνει λοιπόν, η εποπτεία θα διεξάγεται βάσει των συνήθων πρακτικών, σημερινών πρακτικών. Δηλαδή, ε, έχετε εθνικές εποπτικές αρχές στη χώρα προέλευσης και υποδοχής και οι οποίοι συνεργάζονται και δεν αναμένονται αλλαγές σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Ποια είναι η διαφορά ότι τώρα έχετε τις εθνικές αρμόδιες αρχές με τις οποίες συναλλάσσεστε ενώ στο μέλλον θα υπάρχει και η κεντρική εποπτική αρχή. Αλλά νομίζω ότι αυτή θα είναι η μόνη διαφορά. Ε, επαναλαμβάνω την ερώτηση, λέει ο κύριο Σμιτ. Δηλαδή μου απαντήσατε ότι δεν εντοπίζετε εσεί κανένα πρόβλημα με το νέο πλαίσιο για την ανάληψη ταχεία δράση, ξαναλέω, ε, όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όχι. Δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Εάν καταφέρουμε να ε, ιδρύσουμε ένα αποτελεσματικό ενιαίο εποπτικό μηχανισμό δεν βλέπω πρόβλημα. Ακριβώς ένα μέρος της επιτυχίας εκεί βρίσκεται. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δρούμε με ταχύτητα, ανεξαρτησία και ε, ε, έλψη σύγκρουση συμφερόντων. Γι' αυτό το παρόν πλαίσιο ακριβώς είναι προτιμότερο από το προηγούμενο. Σε ό,τι αφορά και με την ταχύτητα πρέπει να το βελτιώσουμε, να είμαστε σε θέση ακριβώς να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις που λαμβάνει το κέντρο με την ίδια ταχύτητα σε εθνικό επίπεδο. Ναι, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ισχυρίζεται κανείς ότι είναι τέλεια ακόμα. Πρέπει να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Πράγμα που θα πράξουμε οπωσδήποτε από τους πρασίνους ο Φιλίπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω την Αγγλική για να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα. Μιλήσατε για τις ασφάλειες, μιλήσατε και για τις τράπεζες. Μία ερώτηση για την καθεμία, για τις ασφάλειες σχετικά με την Omnibus 2, την οδηγία Omnibus 2 και σε σχέση με αυτή την, ε, το ζυγό ε, ε, πτυτικότητας. Η προσπάθεια φαίνεται να μειωθεί αυτή η πτυτικότητα της αγοράς είναι μία από τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι έτσι ώστε να αποφύγουμε τις λεγόμενες fire sales και αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία φούσκας αν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο. Και δεύτερον για τις τράπεζες. Ο συνάδελφος που μίλησε και συμπατριώτης σας είπε στο Βίλνιους ότι υπάρχει πρόοδος στην Ευρώπη, ότι οι τράπεζες τώρα φτάνουν σε ένα ποσοστό μόχλευσης που φτάνει το 3,75%. Ε, κάτι τέτοιο ακούγεται αρκετά ασθενές κατεμέ. Ε, και τι κρίνεται για τις προτάσεις οι οποίες κυκλοφορούν ότι δεν ήμασταν ιδιαίτερα αυστηροί στο θέμα της μόχλευσης και ότι θα έπρεπε να συνδέσουμε το 10% ε, τουλάχιστον για κάποια πιστοτικά ιδρύματα. Πιστεύετε ότι ένας τέτοιος στόχος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθεροποίηση και μείωση ε, της αποφυγής κινδύνων και αποστροφής κινδύνου μάλλον για τις τράπεζες. Για το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε μέτρο το οποίο μειώνει αυτή την επιθετικότητα της αγοράς δεν θα πρέπει να δημιουργεί κίνητρα για υποκεφαλαιοποίηση και αυτό θα δημιουργήσει άλλου είδους κινδύνους, συγκέντρωση κινδύνων και ταυτόχρονα τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμμετρικά στη φύση τους και όχι ασύμμετρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ε, μια ζώνη προστασίας όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν οικονομικά. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι επίσης διαφανή. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι συστηματικά ενήμεροι για τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων. Είναι κάτι το αυτονόητο αυτό και τίποτα δεν θα πρέπει να αποκρύβεται. Αυτονόητο αλλά πρέπει να το λέμε. Για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας. Εμείς ακούσαμε πολλούς αριθμούς δεξιά και αριστερά για το ποιο είναι το σωστό ποσοστό της μόχλευσης. Η Επιτροπή της Βασιλείας είχε πει 3%. Και μετά ακούσαμε το 5% από κάποιους άλλους κύκλους. Όταν κοιτάμε εμείς τα ποσοστά αυτά της μόχλευσης, πρέπει να δούμε ακριβώς και κάποιες διεθνείς συγκρίσεις. Και αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα ποσοστά μόχλευσης είναι χαμηλότερα για τις αμερικανικές τράπεζες από ότι είναι ε, υποχρεωτικά για τις ευρωπαϊκές. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί εδώ γιατί φυσικά υπάρχουν διαφορετικά λογιστικά μέτρα αν εμείς προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας το σύνολο της έκθεσης των πιστοτικών ιδρυμάτων χωρίς το λεγόμενο netting, τότε ε, φοβάμαι ότι τα ποσοστά θα ήταν περίπου τα ίδια ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μας. Το σκεφτόμαστε λοιπόν αυτό το θέμα των ποσοστών μόχλευσης και υπάρχουν πλέον εκτίματα από το να είναι κανείς, με το να είναι κανείς αυστηρός από ότι με το να είναι πιο χαλαρός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι κάποια πολύ αυστηρά επίπεδα μόχλευσης επηρεάζουν τη ρευστότητα. Και ιδιαίτερα ε, τις δραστηριότητες της λεγόμενης χαμηλής απόδοσης οι οποίες πολλές φορές παρέχουν ρευστότητα σε πάρα πολλές ε, αγορές. Αυτό το οποίο πιο συγκεκριμένα κάνουν οι τράπεζες με ένα πολύ δεσμευτικό ποσοστό είναι να ξεφορτωθούν αν θέλετε τις χαμηλής απόδοσης ε, δραστηριότητες, τα ρέπος σαν παράδειγμα. Θα ξεφορτωθούν τα ρέπος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν υπολογίζουμε τις επιπτώσεις των διαφορετικού ποσοστού μόχλευσης για αγορές που είναι απαραίτητες για την νομισματική πολιτική για διάφορους λόγους. Αγορές οι οποίες πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη ρευστότητα και αγορές στις οποίες και το κόστος απόδοσης μερικές φορές είναι ιδιαίτερα χαμηλό και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στα ποσοστά μόχλευσης να καταστρέψουν τις αγορές αυτές και να περιορίσουμε έτσι τις αντισταθμίσεις για πάρα πολλές συναλλαγές. Εμείς το σκεφτόμαστε το θέμα αυτό ακόμα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Όπως πιστέψαμε ε, και πιστεύαμε μέχρι πρόσφατα. Δεν έχουμε λοιπόν μια ξεκάθαρη άποψη για το ποσοστό το 3% της Επιτροπής της Βασιλείας σίγουρα επιτρέπει να υπάρξει μια σαφής αντιμετώπιση των σημερινών πληθωριστικών πιέσεων. Μάλιστα στις Ηνωμένε Πολιτείε επιτρέπεται με κάποιες προϋποθέσεις και χαμηλότερο ποσοστό από 3%. Θα δημοσιεύσετε μια πώληση paper γύρω από αυτό. Όχι, δεν το έχουμε αυτό σαν προοπτική για τον επόμενο χρόνο. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο σκεφτόμαστε και θα το συζητήσουμε και στην επόμενη ε, συνεδρίαση της ε, Διευθυντικής Επιτροπής του Steering Committee. Αν επιτρέπετε να επέμβω εδώ, το Κοινοβούλιο έχει ε, κάποιες επιφυλάξεις, ποσοστώσεις κτλ. Γιατί οι πολιτικοί ε, ασχολούνται με όλα αυτά, με κρατικά ομόλογα, με ε, δάνεια, με υποθήκες και τα λοιπά και όλα αυτά τα βάζουν στην οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει 4. Ε, ε, δεν είναι ακριβώς αυτό στάθμιση κινδύνου. Πάντως όταν θα ασχοληθούμε με την οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει Σκεφτήκαμε ότι η μόχλευση θα πρέπει να είναι διαφορετική ανάλογα με τα διάφορα ε, μοντέλα, ε, τα επιχειρησιακά, επιχειρηματικά και στις τράπεζες η μόχλευση να είναι διαφορετική ανάλογα με τον κλάδο. Αλλιώς, αν είναι κάτι ομοιόμορφο, κινδυνεύει να στραγγαλίσει ε, το σύστημα και είναι κάτι για τεράστια παγκόσμια τράπεζα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι παρόδο για να δείτε πού βρίσκεται η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. Ναι. Μία από τις ε, όμορφες πτυχές ε, του δίκτυ μόχλευσης είναι ότι είναι μια απο τις ομορφες πτυχες του δικτυμου μοχλευσης έννοια που την καταλαβαίνει ο κόσμος. Και δεν χρειάζεται να ε, υπησέρχεται εκεί η στάθμιση κινδύνου. Είναι κάτι σαφές, κάτι εύκολο και αν κατάλαβα καλά αν είχαμε να έχουμε διαφορετικούς δείκτες μόχλευσης για διάφορες δραστηριότητες, ε, χρειάζεται προσοχή εδώ, γιατί καμιά φορά ε, χρειάζεται ένα αρμπιτράζ ε, για να βελτιστοποιηθεί ας πούμε το αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον είναι, αλλά νομίζω ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε την ελκυστικότητα ενός απλού συστήματος, μιας απλής έννοιας που δεν μπαίνει στις επιλογές διαχείριση των τραπεζών. Ο κύριος Φόξ από τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Κύριε Ντράγκη, στις εγωικές παρατηρήσεις σας αναφερθήκατε στη φερεγγιότητα 2 και έχω τρεις ερωτήσεις περί αυτού. Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω πάνω από τέσσερα χρόνια το φάκελο αυτό, οπότε έχουμε μια κοινή επιθυμία. Το αμελητή πρέπει να κλείσει ε, ο φάκελος. Για το νομοθετικό κομμάτι μπορείτε να σχολιάσετε το εξή. Θεωρείτε επιθυμητό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να νομοθετούν λεπτομερώς ή θα προτιμούσατε οι τεχνικές λεπτομέρειες να αποφασίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές και πιο συγκεκριμένα ενδείκνεται για μας να υποδείξουμε εμείς ποσοστά για ορισμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργετικού που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ή πρέπει να επέμβουν καλύτερα οι ρυθμιστικές αρχές και όταν μιλάμε για την νομοθεσία μήπως έτσι δημιουργούμε νέους κινδύνους για το μέλλον δεύτερον. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι κατά τη γνώμη σας που υπάρχουν ε, κατά την εφαρμογή της φερεγγιότητας 2 εάν έχουμε παράπλευρες απώλειες ως προς την χρηματοδότηση για ε, τη χρηματοδότηση των υποδομών. Αυτά μου είπαν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και μήπως αυτό δημιουργήσει ευρύτερο κίνδυνο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τρίτη ερώτηση σε σχέση με την χρήση των ε, αξιολογήσεων επιστοληπτικής ικανότητας. Ε, στην τρίτη οδηγία για τις κεφαλαιοικές απαιτήσει είπαμε ότι για τα credit ratings και για αριθμιστικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σταδιακά να ε, καταργηθούν οι ισχύουσες ε, διατάξεις μέχρι τα τέλη του 2014. Αντίθετα όμως ε, αναφέρονται όλοι, όλα είναι και περισσότερο στην πιστοληπτική ικανότητα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι λογικό αυτό για το Κοινοβούλιο και θεωρείτε ότι συγκεκριμένε αναφορές που υπάρχουν μέσα στη φαραγγιότητα 2 για την πιστοληπτική ικανότητα μήπως μεγενθύνουν το, το, το κίνδυνο, δηλαδή εάν πούμε στους επενδυτές ότι οτιδήποτε είναι κάτω του 3B ε, είναι απαγορευμένο, μήπως έτσι ε, δημιουργήσουμε νέους και μεγαλύτερους κινδύνους για το μέλλον. Απάντηση. Ποιο είναι το βέλτιστο μίξ ανάμεσα στη λεπτομερή νομοτεχνική παρέμβαση και τη διακριτική ευχέρεια των ρυθμιστικών αρχών. Hm. Ε, όχι μόνο για αυτό το ζήτημα, αλλά γενικότερα πιστεύετε ότι εάν η ρυθμιστική αρχή έχει απόλυτη ελευθερία, τότε τελικά έχουμε ρυθμιστικού χαρακτήρα αρμπιτράζ. Εάν είναι άκαμπτη τελείως η νομοθεσία, τότε σε ένα τέτοιο τομέα που υφίσταται διαρκώς αλλαγές, ε, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να είναι απαρχιωμένη η νομοθεσία. Πού τραβάει κανείς τη γραμμή, είναι δύσκολη, δύσκολο ζήτημα. Το θέμα είναι να περιορίσουμε τη διακριτική ευχέρεια τη ρυθμιστική αρχή, ενώ ταυτόχρονα οι νομοθετικέ διατάξει εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν ε, στις ε, ποικίλε, πολλές και ποικίλε περιστάσεις. Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς ακολουθούμε, και να μην το ξεχνάμε αυτό, ακολουθούμε τον εξή δρόμο. Επιδιώκουμε πιο ομοιόμορφα, εναρμονισμένα συστήματα. Οπότε το να υιοθετήσουμε με διαφορετική συμπεριφορά μόνο και μόνο για τη φαρεγγιότητα δύο αυτό θα αντέβαινε στην ε, συνολικότερη ε, νομοθετική τάση των τελευταίων ετών. Δεύτερον, εάν τώρα η φερεγγιότητα δύο μας είπατε μειώνει την ικανότητα των ασφαλιστικών εταιριών για να προσφέρουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στην οικονομία. Ε, δεν έχουμε τεκμήρια προς αυτή την κατεύθυνση προς το παρόν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν μεσομακροπρόθεσμες επενδυτικές πολιτικές οι οποίες διέπονται από την ανάγκη να υπάρχει αντιστοίχηση το, της ορίμανσης των στοιχείων του ανεργητικού με τις ίδιες τις επενδύσεις και πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και μόνο τότε συνεχίζεται η επενδυτική πολιτική. Οπότε Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται τέτοια επιχειρήματα στις συζητήσεις που γίνονται για το πακέτο των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων για τις παραχωρήσεις ανακούφισης, πιστοτικής ανακούφισης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λαμβάνετε και αυτό υπόψη όταν εκτιμάτε την κατάσταση. Επίσης, Κάποιοι πιστεύουν πως ε, τα βάρη κινδύνων πρέπει να αναλαμβάνονται και ο Ιώπα νομίζω έχει δώσει... Α, συγγνώμη, ποια ήταν η ερώτησή σας, όχι, για την πιστοληπτική ικανότητα σας είπα. Είναι ε, σοφό στη φερεγγιότητα 2 να μιλάμε για πιστοληπτική ικανότητα, ενώ στην CRA 3 μόλις ζητήσαμε σταδιακά να εκλείψει αυτό. Γιατί είναι συνετό να ε, γίνεται η μνήα στη νέα νομοθεσία απάντηση. Δεν ε, ε, το έχουμε σκεφτεί ακόμη. Θα σας δώσω μία απάντηση μόλις ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτού του σημείου. Στο μεταξύ βάζουμε ένα κατόφλι τριπλού Β που δεν μπορούν πολλοί να το φτάσουν ακόμα ε, αυτή τη στιγμή. Ενδιαφέρον θα είναι να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Από την ΚΟΟ, ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη αντίστοιχη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, δηλαδή πριν από δύο μήνες, σας είχα ρωτήσει για τις εκτιμήσεις σας σχετικά με την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα και επίσης σας είχα ρωτήσει ότι στην περίπτωση που το ποσό των 50 δις που έχει δοθεί για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δεν φτάνει, τι θα γίνει. Πέρασαν δύο μήνε, δεν θέλω να σα κουράσω με άλλη ερώτηση, επαναλαμβάνω την ίδια ερώτηση, διότι τότε είχατε πει ότι ανησυχείτε κι εσεί με την πορεία που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια, αλλά δεν είσαστε ενημερωμένο για την υγεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματο. Σα ερωτώ λοιπόν, έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω σχετικά με την πορεία των δανείων αυτών. Δεύτερο που έχει σχέση με την ιδιότητά σας, το ύψος των κόκκινων δανείων στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών και βεβαίως και άλλων χωρών. Θεωρείτε ότι αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ελλάδα, άλλη χώρα για την Ευρωζώνη. Και τέλος, αν ο έλεγχος που γίνεται τώρα στις ελληνικές τράπεζες, στους ολογισμούς, από την Τράπεζα της Ελλάδας και την BlackRock, δείξει ότι το 50 δις δεν φτάνει. Τι σενάρια έχετε, τι σκεφτόσαστε, πώς θα το λύσετε αυτό το πρόβλημα, ε, πώς θα γίνει η διάσωση των τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ. Well, we... Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ ε, ακριβώς αυτό το θέμα των δανείων στο Συμβούλιο μας ε, συστημικού κίνδυνου. Δεν είμαστε σε μια στιγμή που μπορούμε να συζητήσουμε και μελλοντικές ε, ανάγκες χρηματοδότηση για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα τελειώνει το 2014, τα τέλη, ενώ του δούνου του μέχρι το 2016. Δεν είναι ακόμα η ώρα να πούμε τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα χρήματα για τα ειδικά θέματα, τα ειδικά δάνεια αυτά δεν το έχουμε συζητήσει όπως σας είπα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Με ρωτήσατε και για την εποπτεία της τραπέζης της Ελλάδος. Θα μπορούσατε ενδεχομένω να επαναλάβετε την ερώτηση σας παρακαλώ. Πολύ ευχαριστώ. Καταλαβαίνω και η κούραση και η διάρκεια της συνεδρίας. Λέω, στην περίπτωση που η έλεγχη που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας, δηλαδή το μέλος σας, έτσι δεν είναι, Ω Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, με αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στου ισολογισμού των ελληνικών τραπεζών. Αντίστοιχο έλεγχο κάνει και η BlackRock. Και φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα να, να ανακεφαλαιοποιηθούν αυτά με τα 50 δι που έχουν δοθεί. Το ερώτημα είναι τι γίνεται, τι σα εισηγείτε, τι κουβεριάζετε με την Τράπεζα τη Ελλάδα αν κουβεριάζετε αυτό το θέμα. No, the present time... Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα αυτό το πρόβλημα. Και όπως σας είπα, το τι μέλη γενέστε θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή οι πόροι είναι αρκετοί, όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Right, thank you. Ωραία, σας ευχαριστώ. Από το Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Λάγκεν. Κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι βέβαιος ότι σας κατάλαβα καλά ε, ως προς τα ταμεία ε, παροχής χρημάτων, το funding και την, ε, τις παρατράπεζες και τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς συμφωνείτε με αυτό που προτείνει το Συμβούλιο να απαγορευτούν αυτά που, που έχουν ε, κάποια κειμενόμενη λειτουργία περισσότερο προτιμάται παρά ένα 3 ή 5%. Επίσης, τα CCPs ε, που κάνουν το clearing ε, για τα παράγωγα βλέπουμε ποια είναι η αγορά παγκοσμίω για τους αντισυμβαλωμένους. Είπατε το netting ότι είναι πολύ πιο επισφαλές ή Μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι για τα CCP. Αν θυμάμαι καλά, το 15 Σεπτεμβρίου του 8, 1,27% κίνδυνο κίνδυνος ήταν ε, από ισολογισμούς ε, των Αμερικανικών τραπεζών, ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η διασύνδεση, αυτό το netting, ε, και είπαμε ότι θέλουμε από κοινού να δράσουμε και εσείς ε, είπατε ότι η ΕΣΜΑ που είναι η αρμόδια αρχή κάνει τώρα τις προτάσεις. Ε, τι γίνεται ε, όμως με το clearing που χρησιμοποιούν τα παράγωγα οι εταιρείε για να εξασφαλίσουν επενδύσεις ή αγορές. Αυτό εσείς πώς το αξιολογείτε. Και η τρίτη ερώτηση έχει γίνει ήδη συνεργασία με την Επιτροπή της Βασιλείας. για την αξιολόγηση μηδενικού κινδύνου ε, ε, όταν πρόκειται για κρατικά ομόλογα. Επειδή συμμετέχετε και εσείς σε αυτές τις δραστηριότητες, είναι δυνατόν μακροπρόθεσμα αυτή η αξιολόγηση κινδύνου για κρατικά ομόλογα μηδενικού κινδύνου σιγά σιγά να ευθυγραμμιστεί με την πραγματικότητα και με τη ρεαλιστική θεώρηση για να ξεπεράσουμε έτσι, μακροπρόθεσμα κάποια από τα προβλήματα που σήμερα έχουμε. Ευχαριστώ. Thank you. The, well, Ευχαριστώ. Ε, Εγώ είπα ότι για τις ε, χρηματαγορές ό,τι είχα να σας πω πριν. Νομίζουμε ότι τα λεγόμενα σύναυς θα πρέπει να ε, περνούν από τις ίδιες προβλέψεις ε, με τις τράπεζες και πρέπει ακριβώς ε, να οδηγηθούν στην λεγόμενη κατηγορία βίναυς. Ε, σας είπα ότι είχα να πω. Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης όπως είπε και η πρόεδρος μας σε σχέση με την αρχική πρόταση. Για τα παράγωγα τώρα. Μία από τις καλύτερες εξελίξεις στα πλαίσια των προσπαθειών που έγιναν για να βγούμε από την χρηματοπιστωτική κρίση είναι ότι όλα τα λεγόμενα standard derivatives και όλες οι συμβάσεις παραγόνων εκαθαρίζονται μέσω των CCP και τα δεδομένα θα φυλάσσονται ε, στα αποθετήρια. Για τα μη standard παράγωγα θα υπάρχει διαφορετική διαδικασία clearing η οποία όμως θα εμπεριέχει πιο θα έλεγα τιμωρητικές, πιο κυρωτικές απαιτήσεις σε επίπεδο κεφαλαίου. Η διαδικασία συνεχίζεται όπως σας είπα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι περιμέναμε όλοι και εσείς μάλιστα γιατί ήσασταν και ο εισηγητής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν στο θέμα των παραγόγων να εργαζόμεθα από δύο γωνίες. Πρώτον, μέγιστη δυνατή διαφάνεια από τη μία και από την άλλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των CCP. Τα CCP μπορεί να καταστούν πηγή συστημικού κινδύνου. Uh, Τα μη ομοιοποιημένα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα συνολικά στην Ευρώπη, θα μεταφέρονται στις εθνικές εποπτικές αρχές το ίσμα και το SRB βέβαια. Αυτό θα επιτρέψει τη μελέτη των, τύπων της έκθεσης και των συγκεντρώσεων αυτού του είδους των παραγωγών. Το SRB έχει σαν στόχο να κάνει συστάσεις σε όλες τις εποπτικές αρχές σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο και να δημιουργήσει ένα φόρουμ διαλόγου επλέκοντας όλες αυτές τις αρχές σε μόνιμη βάση. Το SRB όπως γνωρίζετε καλά, θα του ζητηθεί στα πλαίσια του ΕΜΗΡ να δώσει και μακροπροληπτικές απόψεις σε σχέση με την διαλειτουργικότητα, όπως είπα στην εισαγωγική μου παρουσίαση. Very difficult question on... Uh, Για το πάρα πολύ δύσκολο θέμα της στάθμισης των κινδύνων. Last General Meeting. Στα, πλαίσια της τελευταίας συνάντησης της διοίκησης της τράπεζας στις 19 Σεπτεμβρίου μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και πανεπιστημιακών παρουσίασαν μια τεχνική έκθεση για το θέμα αυτό και στο, προς το Συμβούλιο του SRB. Έχουμε μπροστά μας να κάνουμε μια πολύ πλούσια συζήτηση. Ήταν μέχρι τώρα καποφόρα είναι ένα σημείο εκκίνησης η έκθεση αυτή έτσι ώστε να αξιολογήσουμε σωστά την έκθεση που δημιουργεί το δημόσιο χρέος και πώς μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος που δημιουργείται. Αλλά δεν προβλέπεται συγκεκριμένη πολιτική πρόταση σε σχέση με την τεχνική έκθεση. Ούτε δεν υπάρχει προειδοποίηση που να προβλέπεται στα πλαίσια του SRB, ούτε σύσταση καν. Θα συνεχίσουμε όμως την προσπάθεια που ξεκινήσαμε, θέλοντας να δημοσιεύσουμε μία έκθεση επιστημονικής φύσεως. και θα σας ενημερώσω όταν υπάρξει μια κάποια πρόοδος σε εύθετο χρόνο. Ταυτόχρονα περιμένω ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί πριν από την αξιολόγηση και τα stress test τα οποία θα κληθεί να κάνει το SSM. Αυτό. Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ώρα τα Υποκρίσεις τρεις ώρες σας έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την πληροφόρηση. see Και στο επανειδήν και σύντομα να μας ξανάρθετε. So that's it until tomorrow at 9.